Καθίστε για να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση όπου θα μιλήσουμε για την ε, καινοτομία, την ανάπτυξη και το μέλλον της ε, διεθνούς συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κορυφαίους καλεσμένους, θα σας τους συστήσω εντός ολίγου και φυσικά και δύο ιδιαίτερους καλεσμένους αργότερα, την είπατε εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη και τον Bill Gates που θα έρθουν αργότερα, γύρω στις 4, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα, την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Think Tank που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση σήμερα, γιατί πραγματικά η στιγμή είναι πολύ επίκαιρη. Φτάνει στο τζακ αυτή η συνεδρίαση. Τώρα που ξεκινάμε τη συζήτηση για τον επόμενο γύρο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα περίοδο προγραμματισμού για το πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανίσει τα αναπτυξιακά της κονδύλια στο μέλλον. Και όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα αυτό, το νέο πρόγραμμα, θα το διαπραγματευτούν οι Υπουργοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει θέσει επιτάπητος και οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν ως νούπο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μορφή που θα λάβει. Έχουμε μια νέα πρόταση που συγχωνεύει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της αναπτυξιακής συνεργασίας σε ένα ενιαίο μηχανισμό. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη διορίσει του εισηγητέ του. Ένα από αυτού είναι στο πάνελ, ο κύριο Γκιόρεν. είναι ένα από του εισηγητέ τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Έχουμε και τον Φρανκ Έγκελ, το δεύτερο εισηγητή τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Και επίση έχουμε κοινή νομοθετική αρμοδιότητα με την Επιτροπή Εξωτερικών. Για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνεργασία των δύο επιτροπών, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, και των συνεισηγητών του που από κοινού θα πρέπει να καταλήξουν για το πώ ε, θα δαπανώνται τα αναπτυξιακά κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλέ είναι οι και τα ζητήματα που θα εξετάσουμε. Βέβαια όλοι συμφωνούμε στην Επιτροπή ανάπτυξη, αλλά και γενικώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ε, υλοποιήσει του στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης, το σύνολο του ΠΔΠ, εσωτερικούς και εξωτερικούς δηλαδή στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να χρηματοδοτούν το θεματολόγιο του 2030. Οπότε είναι πολύ έγκαιρη αυτή η διοργάνωση και μάλιστα μερικοί ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία είναι παρόντες και θα ακούσουμε προσοχή την άποψη των think tanks αυτών των ομάδων προβληματισμού και την άποψή τους ως προς τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς ε, ε, θα, δι... θα διαμορφωθεί η ανάπτυξη στο μέλλον. Σάιμον, μπορείς να μας παρουσιάσει το πρώτο πάνελ. Καταρχήν σας ευχαριστώ που βοηθήσατε στη διοργάνωση. Ήσασταν πραγματικά πρωταγωνιστές, τη, πρωταγωνίστρια της ε, Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και ως πρόεδρος της ΔΕΒΕ και πέραν ε, αυτού. Μακάρι να συνεχίσετε σε δύο-τρει ακόμη κοινοβουλευτικές θητείες για να συνεχίσετε το πολύ αξιόλογο έργο σας. Είμαστε ευγνώμονες αυτό που κάνετε. Ε, την αποκαλούμε έκτακτη αυτή τη συνεδρίαση, γιατί ε, ε δεν θα ε, ξοδέψουμε άλλες 4-5 ώρες για να συζητούμε το Brexit. Αν έχει κανείς λύση για το μηχανισμό ασφαλείας για τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία, το backstop δηλαδή, γράψτε το σε ένα χαρτά και στείλτε το στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όμως ένα περίπλοκο πρόγραμμα το απόγευμα. Θα σας εξηγήσω πώς θα εξελιχθεί. Καταρχήν, λίγο πριν τις 4, έχουμε μία συζήτηση ε, δημαρχείο θα έλεγα. Δηλαδή όχι μια κλασική συζήτηση ε, εμπειρογνωμόνων. Θα δώσω το λόγο στην Ομίγυρη και μετά θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και θα ήθελα να σας θέσω τα ζητήματα που θα συζητήσουμε και θέλω να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Μετά ίσως γίνει κανένα δίλεπτο διάλειμμα και στις 4 περιμένουμε τη Φεντερίκα Μογκερίνη και τον Bill Gates. Θα μας μιλήσουν και οι δύο και μάλιστα ε, και με Σόλτς. Ε, θα κάνει σχόλιο από το Ομονικό Ινστιτούτο και φυσικά θα γίνει συζήτηση με τους ναι. ευρωβουλευτές. Και θα ολοκληρώσουμε με συμπεράσματα. Ε, πρέπει να φύγω λίγο πριν τις 5 γιατί ε, αναζητούσαν μανιωδώς χρόνο για διμερή, διμερή επαφή και βρήκαν μόνο γύρω στι 5. Γι' αυτό θα τελειώσουμε ίσω και 10 λεπτά νωρίτερα. Και επίση θα έχουμε εκτό από τον Φρανκ Έγκελ, τον James Μάκη, διευθυντή του Ινστιτούτου του Μάστρικ και τον Ζεμπαστά Τρεγέρ, πρόγραμμα, διευθυντή προγραμμάτων στην ομάδα εργασίας μας. Ε, μεταδιδόμαστε και από το διαδίκτυο, οπότε αν είστε διακριτικοί και ταυτόχρονα μπορείτε να είστε και προκλητικοί. Πάντως η ιστορία θα μας κρίνει, μας καταγράφει. Επίσης έχουμε και ένα hashtag στο Twitter, το hashtag ETTG2018. Ίσως είναι χρήσιμο να συνεχιστεί η συζήτηση και μέσω Twitter στη διάρκεια της ε, ε, διάσκεψής μας. Έχουμε πραγματικά κορυφαίους ε, καλεσμένους και, στη, και στην, στο πάνελ και στην ομιγύρη. Νάταλη Τότσι είναι ε, σημαντικός παράγων και στηρίζει την εξωτερική στρατηγική της Φεντερίκα Μαγκερίνη. Ο Άλεξ Τιερ είναι ε, εκτελεστικός διευθυντής του ODI του Ινστιτούτου στο Λονδίνο, από τους σημαντικότερους, ε, από τους σημαντικότερους μηχανισμούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Η Άννε Μπυργίτε Άλμπερτσεν, διευθύντρια του Plan International τον Αντεμπάιο Ολουκοσί, που είναι διευθυντή για την Αφρικα και τη Δυτική Ασία στο Διεθνέ Ινστιτούτο Δημοκρατίας και Εκλογική ε, Αρρωγής και πρόεδρο ε, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου του ECDPM και τον Άλεξ Τιερ από το Λουξεμβούργο. είναι το, ποιο είναι το κυρίως θέμα και να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις πριν ξεκινήσουμε. Επίσης, αν κάποιοι ευρωβουλευτές κάθονται ε, πίσω, μπορούν να προχωρήσουν τα μπροστινά καθίσματα. Αν αρχίσει να φαίνεται ότι εκνευρίζεται, ίσως πρέπει να απομακρυνθεί πάλι. Αλλά αν μετακινήσετε μπορεί να χάσετε και τη θέση σας. Του χρόνου έχουμε εκλογές και έχουμε μεγάλες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε ε, Spitzenkandidaten, ε, επικεφαλής ψηφοδελτίου για τη θέση του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό μέχρι το 2027. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική συγκυρία για τη διαμόρφωση του μέλλοντο. Και είμαι πολύ περίεργο και ίσω μα βοηθήσουν εδώ οι ευρωβουλευτές ε, να καταλάβουμε ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το θέμα τη διεθνού συνεργασία. Υπάρχει συνένεση ή υπάρχουν απόψεις ε, ιδεολογικές γενικώ για το ποιο είναι ο δικαιούχο τη ενίσχυση, πώ δαπανάτε, πώ συνδυάζεται με την ανθρωπιστική βοήθεια, τι γίνεται με το εμπόριο, το κλίμα, την ασφάλεια, τη μετανάστευση. Σε μερικέ χώρε δεν γίνεται καν συζήτηση γιατί όλοι συμφωνούν. Σε άλλε χώρε όμω υπάρχουν σοβαρέ διαφωνίε. Θέλουμε να μάθουμε αυτέ τι διαφορέ. Εκεί που α, ε, δεν υπάρχει διαφωνία είναι για τι θεμελιώδει αρχέ. Και πριν α, ε, ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σα δοκιμάσω ε, με κάνουμε δύο ψηφοφορίες. Σκεφτείτε λοιπόν το εξή. Θέλω να ψηφίσετε ναι, όχι ή δεν γνωρίζω. Η πρώτη ερώτηση είναι, ο κόσμος είναι τέλειος όσο, το, όσο καλύτερος γινόταν. Ε, σηκώστε το χέρι αν συμφωνείτε ή τώρα σηκώστε το χέρι αν διαφωνείτε. Ε, σηκώστε το χέρι αν απέχετε, αν δεν ξέρετε. Δεν είναι και πολύ. Οπότε δεν είναι και πολύ αυτοί που δεν ξέρουν. Επίσης έχουμε πολύ έργο μπροστά μας. Τώρα, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξη για το 2030 είναι μια καλή περιγραφή για το πού θέλουμε να φτάσουμε, αλλά όχι αρκετός ή ε, ε, επαρκής οδικό χάρτη για το πώ θα το καταφέρουμε. Έχουμε πολλές πτυχέ τη βιώσιμη ανάπτυξη. φτώχεια, βιωσιμότητα και το άλλο ποιο είναι, α, η συμμετοχή. Ποιο είναι, ε, είναι υπέρ των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, Ποιο είναι κατά. Α, ένας είναι κατά. Καλά, θα μας τα πείτε αργότερα. Πολύ καλός προορισμός η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά κακός δικός χάρτης, χάρτης πορείας. Ε, φυσικά όλοι ενδιαφερόμαστε για τη φτώχεια. Ξέρουμε ότι ο κόσμος πάει χάλια, ε, η πολυμέρεια απειλείται και διαβρώνεται και η παγκόσμια τάξη. Ω προ αυτά συμφωνούμε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για όλα αυτά. Τι εναλλακτικέ προτείνουμε για να λύσουμε την κρίση. Και ιδιαίτερα για μας στην Ευρώπη. Γιατί εδώ μιλούμε για το μέλλον της, Ευρω... της Διεθνούς Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά και τι δεν μπορεί να κάνει. Οι πέντε διευθυντές ε, της ομάδας μας δημοσίευσαν ένα άρθρο στο Euractiv και όλοι λέμε ότι η αυτόματη απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα του κόσμου δεν είναι η Ευρώπη. Πολύ συχνά η σωστή απάντηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα στον κόσμο είναι η Ευρώπη, αλλά όχι πάντα. Οπότε εμείς θα διακρίνουμε πού ε, έγκυται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού μπορούν 28-27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνεργασία τους να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και τι πράγματα θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρο και να πούμε αυτά είναι για άλλους. Αυτά είναι τα πιο, βασικά, τα πιο βασικά θέματα. Ποια είναι τα πιο κατεπήγοντα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο κόσμο, όχι κανένα μακροσκελή κατάλογο. Και τι, το δεύτερο ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες, ε, ε, η διαδικαστική είναι εξή. Σεβόμαστε τους ευρωβουλευτέ, σίγουρα θα του δώσουμε το λόγο, αλλά παρακαλώ όλους ε, να σηκώνουν το χέρι αν θέλουν να μιλήσουν και να μιλάνε το πολύ για 1,5 λεπτό. 75 με 90 δευτερόλεπτα. Πείτε ποιο είστε, πείτε κάτι ενδιαφέρον και μετά από 90 δευτερόλεπτα βάλτε τελεία. Γιατί θέλουμε ανταλλαγή απόψεων, διάλογο και ερωταπαντήσεις, όχι λογίδρια και διαλέξεις. Και μετά θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες για να μας παρουσιάσουν τη δική τους κόπια. Πάντως, είναι συνεδρίαση, διάλογος και όχι παρουσίαση των ομιλιών των εμπειρογνωμών. Οπότε σηκώστε το χέρι ποιος θέλει το λόγο πρώτος. Η Λίντα λέει και είναι το αφεντικό. Όσοι κάθονται πίσω έρθουν πιο μπροστά, έστω και στις θέσεις των Ευρωβουλευτών. Οπότε, ποιος από την Ομίγυρη θέλει το λόγο. Ε, γιατί να μιλήσει ο κύριος που είναι κατά των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και μια ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων ή μεταξύ των γενεών. Δεν θα μιλήσει κανείς άνω των 60. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάπως ε, έχουμε κουραστεί να πρασπιζόμαστε εμείς τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα έπρεπε να είμαστε οι μόνοι. Γι' αυτό λοιπόν ε, προ ε, την επόμενη θητεία πρέπει να εστιάσετε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η πρόκληση. What would you do differently? Τι θα κάνετε διαφορετικά ή τι θα έπρεπε να κάνουν διαφορετικά οι ευρωβουλευτές απάντηση. Θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο ε, στην αναβάθμιση ε, της κατάστασης, ε, όπως παραδείγματο χάρη για την Πολωνία και την Ουγγαρία, κάποια πράγματα που συμβαίνουν, η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και δι των γενικών πρέπει να αυξηθεί. Τι γίνεται με αυτούς που δεν πληρούν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέλος πάντων. My name is Κάρολ Uitendale, λέγομαι από το Βέλγιο και συμμετέχω στο πρόγραμμα κύκλος κινητικότητας των νεαρών Αφρικανών επαγγελματιών. Έχουν σπουδάσει και εκεί έχουν το υπόβαθρο το αφρικανικό, έρχονται για ένα χρόνο εργάζονται εδώ και πηγαίνουν πίσω στις χώρες τους. Εγώ θα απευθύνω έκκληση για την εκβιομηχάνηση τη Αφρική. Αυτή είναι η λύση, κατά την άποψή μου. Να δώσουμε κίνητρα σε δυτικού επιχειρηματίε να πάνε να επενδύσουν στι ε, επιχειρηματικέ βιομηχανικέ δραστηριότητε στην Αφρική. Μιλάμε για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά ε, ξεχνάμε ότι είναι και προ το δικό μα όφελο να επενδύσουμε στην Αφρική. The academics are talking about deindustrialization or Ξέρετε, πολλοί μιλάνε όμως για πρόορη αποβιομηχάνηση ή ε, αποβιομηχάνηση στην Αφρική. Ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Κάποιος άλλος θα ήθελα να πει τίποτα εκεί δύο στο βάθος παρακαλώ και οι δυο σας θα λάβετε το λόγο. Ορίστε. Γεια σας. Mary Aikenbrook λέγομαι. Είμαι ασκούμενη στη ΔΕΛΤΑ ΕΞΠΟ για τις εθνείς σχέσεις. Είμαι από τις Ηνωμένε Πολιτείε, το καταλαβαίνετε από την προφορά μου ίσως, αλλά αυτή με έφερε στην Ευρώπη αρχικά. Ήταν ε, ένα πρόγραμμα του Erasmus Mundus ε, που μου άλλαξε τη ζωή πραγματικά. Ήταν ε, τόσοι πολλοί αυτοί που γνώρισα, που είχαν έρθει για, στο πλαίσιο των σπουδών τους και άλλαξαν όμως κατεύθυνση και γύρισαν στις χώρες τους και Εντάξει, μπορεί στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, να μην έχουμε το ίδια πλεονεκτήματα, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οργανώσει υποτροφίε, βοηθούν ε, τον κόσμο στις χώρες τους. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε προγράμματα που χώρες ε, που δεν είναι τόσο προηγμένες θα μπορέσουν να βοηθηθούν από την Ευρώπη. Και η κυρία πίσω σας τώρα. Um, good afternoon. My um, Λέξ Γκίμπ λέγομαι από Καμπότζη και Ηνωμένες Πολιτείες, Καμποτζοαμερικάνα. Και εκπροσωπώ τη φωνή της Καμπότζης που έχει συγγύσει εδώ και χρόνια. Και θέλω να μιλήσω για τις εκλογές του 2018 στην Καμπότζη. Η κυβέρνηση έχει μια ωραία ρητορική, τα λέει πολύ ωραία, όμως τα πράγματα έχουν αλλιώς. Ζω πολλά χρόνια στην Αμερική, αλλά δεν καταλείπει την Καμπότζη από τα μυαλό μου και θα πρέπει να ξέρετε ότι η Καμπότζη έχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού που υποφέρει σιωπηλά. Και πρέπει ο κόσμος να ξέρει τον πόν, με συγχωρείτε, συγκινούμε. Και υπάρχει και κάποιος που είναι εδώ σε αυτό το κτίριο και ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει την ανθρωπιά και την αγάπη. Ο Λοράν Καβέν, που είναι ο πρόεδρος του κόμματος κατά της φτώχειας ο πρόεδρος του κινήματος Δικαιοσύνη για την Καμπότζη. Συγγνώμη, θα σας διακόψω γιατί ενώ λέτε πολύ σημαντικά πράγματα έχετε περιβεί δυστυχώ ε, τα 90 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα τώρα το Σαλ Γκέρενς να ζητήσω να κάνει τα σχόλιά του. Δεν μας αρέσουν, μας αρέσουν τελικά οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, δεν τα πάει καλά στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν, έχουν και τις ευρωεκλογές. Ε, για καθοδηγήστε μας παρακαλώ. Je crois que <clears throat> la communauté internationale a déjà répondu à la première. Ήδη έχει ανταποκριθεί σε αυτό το πρώτο που είπατε. Σε αυτό που ρωτήσατε, απάντηση δεν κοινότητα. Ναι, του θέλουμε του στόχου αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι από κύμα διεθνού συνένεση σε επίπεδο ΟΗΕ. Είναι πρόκληση να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι με πολυμερείς μεθόδους όπου να πρωταγωνιστεί βέβαια η Ευρώπη γιατί η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε χαρακτηρίζεται από μια οικοδόμηση διεθνούς ε, ε, διακυβέρνησης ούτως Αλλά γιατί είναι, είμαστε σε κοινωνία μου γιατί έχουμε τον πρόεδρο τον Ήπα που ό,τι έτσι ακόμα και να μοιάζει με πολυμέρεια ε, διότι τι κάνει η Ευρώπη τότε θα πρέπει εκείνη να περισσώσει ό,τι σώζεται σε επίπεδο διεθνών σχέσεων η Ευρώπη να προσπαθήσει να εξαγάγει το πρότυπό της για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ναι. Απειλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. ποτέ δεν είναι κάτι το κεκτημένο, το δεδομένο Εσαί. Ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη που αγνοούν, κάνουν ότι δεν ξέρουν, καταπατούν αυτά που γράφει η συνθήκη. Ξέρετε για ποια κράτη μιλώ. Οπότε θα πρέπει κάπως να μπει ένα τέλος αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να βρεθούν οι μηχανισμοί και ε, να αντιμετωπιστούν αυτοί που φέρνουν τέτοια δυσλειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει έτσι να δούμε πώς θα καταφέρουμε παράλληλα και να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρώπη να είμαστε άψογοι και άπαξ και το καταφέρουμε τότε θα μπορέσουμε να πείσουμε και τους άλλους να εμπνευστούν από το ευρωπαϊκό μοντέλο. Διακόπτει ο πρόεδρος Υπήρξε ποτέ άψογη η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εσείς μας δείτε ότι ε, μόνο εάν είναι άψογη η Ευρώπη άμεμπτη τότε μπορεί να κουνήσει το δάχτυλο στους άλλους. Μα όμως μήπως ε, αυτό είναι μια ψευδέστηση για τις παλιές καλές μέρες. Είναι έτσι. Γκέρενς. γίνει αποδεικτό από την Κίνα, ένας δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας. Οπότε και έτσι να υπάρχει ένα ενδικό μέσο για αυτούς που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στον πρώτο βαθμό. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπει στα πρώτα σέλιδα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο θα είμαστε περήφανοι. Ενθαρρύνει η Ευρώπη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θεμελιώδης αρχή που ενσωματώνεται στις συνθήκες. Οπότε, αυτοί που γιορθώνουν τα κακό τους, τους, έχουν τις βοηθειάς μας. Οι συνομιλητές μας να είναι κράτη που πολλές φορές σχετίζονται με κυκλώματα διαφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε πώς θα κόψουμε τα φτερά αυτόν που πρέπει. Κάνει όμως ότι μπορεί η Ευρώπη, έχουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τι πρωτοβουλίε. Αυτό είναι σημαία μα ως πρωτοβουλία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με άλλου τρεις συνεισηγητέ. Εδώ έχουμε τον κύριο Έγκελ, εξ αυτών, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να μπορέσουμε με αυτή την υπόθεση να αποκτήσει αξιοπιστία αλλά και αποφασιστικότητα η Ένωση. Μάλιστα, βαθμία προσέγγιση. Βήμα, βήμα. Κυρία Χιμένος, Ευρωβουλευτή. Να σας τα πω στην μητρική μου γλώσσα. Ακριβώς πάνω σε αυτό που ρωτήσατε, αν μας αρέσουν ή όχι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ναι, ναι, σήκωσα το χέρι μου. Σας είπα ότι μου αρέσουν. Έχουμε το 16 που αφορά την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και θωρακισμένους θεσμούς. Αυτά είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης. Χωρίς ασφάλεια δεν έχουμε επενδύσεις, χωρίς επενδύσεις δεν έχουμε εκβιομηχάνηση και δεν έχουμε άρα και ανάπτυξη, τελικά δεν έχουμε δουλειά. Μιλάμε τώρα ε, για καινοτομία. δεν ξέρω αν υπάρχει όμως η ασφάλεια. Να μην έχουμε προκαταλήψει ιδεολογικές όταν έρχεται η ώρα διάθεσης πόρων στο α, στο β, β μέρος το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συστρατευτούμε για την ασφάλεια ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχει απασχόληση και ε, στρατηγικός στόχος δυο ανάπτυξης της χιλιετίας είναι η συμμετοχή, η χειραφέτηση των γυναικών. και εδώ να μπει η καινοτομία. Και επίσης έχουμε και στον φορέα πλάν ε, διάφορες προτάσεις ε, από πλευράς ε, ηλιακής ενέργειας και άλλα τα οποία θα μπορούσαν να εμπλέξουν τις γυναίκες. Αυτές θα πρέπει να εμπλακούν και έτσι να πάμε στην ανάπτυξη που θέλουμε. Τι, γιατί είναι ασφάλεια. επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση στα αγγλικά. Ίσως η προσέγγιση έχει κάποιες συνέπειες ε, ε, στη χρήση των κονδύλιων του προπολογισμού. Δηλαδή, ε, θα πρέπει κάποια κονδύλια να μεταφερθούν από το νέο ενιαίο χρηματοδοτικό όργανο μέσω μηχανισμό και να μπει στο, στο μηχανισμό για την ειρήνη ή να μεταφερθεί κονδύλια από ορισμένες χώρες σε άλλες, γιατί σίγουρα συνέχεια δημιουργούνται νέα ταμεία, αφαιρούνται κονδύλια από τα αναπτυξιακά υπουργεία και μεταφέρονται στα αμυντικά υπουργεία και ούτω καθεξής. Ε, δεν είμαι ειδήμων στα θέματα ασφάλειας και δεν λέω ότι θα πρέπει, από πού θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κονδύλια και πού θα πρέπει να μεταφερθούν. Αλλά όταν μιλούμε για τη μετανάστευση, γιατί εγώ κατάγομαι από την Ισπανία, από την Ανταλουσία και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Όλοι μιλάνε για το σχέδιο Marshall, αλλά κανένας δεν λέει πώς θα το εφαρμόσουμε. Στις ιδέες καλά τα πάμε, αλλά δεν υπάρχει περιεχόμενο. ίσως αμέσω απευθείας από τις χώρες ίσως. Και όταν μιλούμε για κονδύλια, για τη συνεργασία, πολλές φορές ακούμε είναι πολύ αόριστα όλα αυτά, δεν ξέρουμε πραγματικά πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Αν τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά, για παράδειγμα για την Ισπανία, είναι πολύ σημαντικό για να σταματήσουμε τη μετανάστευση, να προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το μεταναστευτικό φαινόμενο Ίσως θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ μεθόδους και να μην τα συγκεντρώνουμε όλα σε ένα ενιαίο ταμείο, αλλά σε διαφορετικούς τομείς όπου τα κράτη ε, θα μπορούσαν να δραστηριοποιούνται περισσότερο στο α ή β σχέδιο. Ε, ας ε, αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο στην ασφάλεια και πώς συνδυάζεται με την αναπτυξιακή ε, βοήθεια, γιατί εσείς ασχολείστε με τα θέματα αυτά. Ναι, Υπάρχει εδώ πρόβλημα όντως μεταξύ θεωρίας και πράξης. Στη θεωρία όλοι συμφωνούμε ότι χαιρόμαστε που έχουμε το στόχο 16 της βιώσιμης ανάπτυξης και χαιρόμαστε που έχουμε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και σίγουρα η ασφάλεια είναι ε, κέριο σημείο, κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης, στη θεωρία τουλάχιστον. Το θέμα είναι στην πράξη πώς θα εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι και πώς εφαρμόζονται ήδη αυτοί οι στόχοι στην πράξη. Γιατί αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι καταρχήν αντί α, να ξεκινάμε και να διευρύνουμε την ασφάλεια για να περιλάβει αν και την ενέργεια και την απασχόληση και το κλίμα και την ασφάλεια και ένα σωρό άλλα θέματα, τελικά στην εφαρμογή ακριβώς επειδή ε, ανησυχούν οι κοινωνίες μας, έχουν βάσιμους αφενός φόβους και αφετέρου ενδίδουν στην κινδυνολογία των λακιστικών κομμάτων, τελικά μειώνουμε τα κονδύλια της εφαρμογής. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Τι εννοούμε. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις ε, στην ανάπτυξη ή θέλουμε μια μεταστροφή των επενδύσεων από τη μία προτεραιότητα στην άλλη. Και ομάδα σαν τη δική μας, την ETTG, είμαστε ε, ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε το στόχο 16. Αυτό που μας ε, ανησυχεί είναι η συρρήκνωσή του και θα θέλαμε αύξηση των επενδύσεων στην εξωτερική πολιτική και στην ανάπτυξη γενικώ. Άλεξ, ήσουν από τους ε, αρχιτέκτονες των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην προηγούμενη σου θέση. Μπορείς να συνεχίσεις εσύ να απαντήσεις αυτήν την ερώτηση. Ναι, σίγουρα. Καλούμαστε να κάνουμε μια πολύ κρίσιμη, να λάβουμε μια πολύ κρίσιμη απόφαση και επιλογή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πώς θα κατανείμουμε τους σπόρους. Γιατί, ναι, με συμφωνώ ότι ο δικός χάρτης για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι πλήρης, αλλά ήδη έχουμε κάποια στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να εξαλείψουμε την εξαθλίωση, την ακραία φτώχεια μέχρι το 2030. Και ξέρουμε που θα εντοπίζεται η ακραία φτώχεια, κυρίως σε χώρες ε, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτε, ε, έχουν ένοπλες ε, σειράξεις. Και γνωρίζουμε ότι οι πόροι γενικώ, συμπεριλαμβανομένα και το πόρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατευθύνονται επαρκώ σε εκείνε τι χώρε, σε εκείνου του λαού που χρειάζεται να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια, από την εξαθλίωση. Και ο μόνο τρόπο να υλοποιήσουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη είναι να επικεντρωθούμε πρώτα στου φτωχότερου. Γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε να αφήσουμε κανέναν πίσω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτού ε, αφού έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα, αλλά πρώτα να βοηθήσουμε τον κόσμο να, καλύψει το χαμένο έδαφο. Επίση, να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε όλων αυτών για την ευρωπαϊκή ε, πολιτική για την παροχή αρρωγής και να επικεντρώσουμε τη βοήθεια στις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να επικεντρώσουμε τους πόρους ε, στις πιο ευάλωτες χώρες. Και αυτό είναι θέμα στόχου 16. Γιατί μερικές χώρες είναι ευάλωτες όχι μόνο επειδή είναι φτωχέ, αλλά επειδή υπάρχει αποκλεισμό, υπάρχουν προκλήσεις στη διακυβέρνηση, υπάρχει ε, μεγάλη περιθωριοποίηση και διακρίσεις μεγάλες. Θα πρέπει λοιπόν ο αναπτυξιακός περιπολογισμό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καλό θα να προωθήσει αυτέ τις προτεραιότητες. Αυτό προβλέπει χάρτα και εκεί θα έχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και αν ε, θέλουμε να ευοδοθούν ε, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό δεν θα επιτευχθεί μόνο χάρη στην παγκόσμια κινητοποίηση, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρωτοστατήσει για να επικεντρωθούμε σε αυτό όταν οι υπόλοιποι ε, δεν το κάνουν. Όντως, αυτή είναι τεράστια πρόκληση για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και τον τομέα 6 της αναπτυξιακής συνεργασίας. Γιατί αν επικεντρωθούμε σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις χώρες που μαστίζονται από ένα σειράξεις, όπως είπε και η Τερέζα, να βοηθήσουμε ε, τους παραδοσιακούς πόρους, αλλά να είμαστε ρεαλιστές για το αν υπάρχουν και να, να δούμε ε, ποιες, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και δεύτερη χώρα δικαιούχος από τις μεγαλύτερες, από τις 10 που λαμβάνουν την ενίσχυση, είναι η Τουρκία. σε πίσω, 90 δευτερόλεπτα, να πείτε και ποια είστε. Τζάκλι Χέιλ από το Save the Children στην προσφώνησή του προ το Κοινοβούλιο με θέμα την ε, κατάσταση και το, ε, της Ευρώπης μίλησε για την Αφρική και είπε δεν χρειάζεται πλέον φιλανθρωπία. Συμφωνείτε προς τα μέλη του ΠΑΝ, ε, ως προς την εξίσωση αυτή βοήθεια ε, με φιλανθρωπία. Ποια θέση θα έχει η βοήθεια στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης της Ένωσης στο μέλλον και κάτι σχετικό. Η μετατόπιση προσεγγιμένε επενδύσει του ιδιωτικού τομέα συνάδει με του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα φτάσει στο στόχο τη αυτή η βοήθεια. Θα ήθελα να ακούσω τι απαντήσει των μελών του πάνελ. Θα ακούσουμε του υπόλοιπου του πάνελ σε λίγο. Αλλά θέλω εσεί να μου πείτε τι πιστεύετε. Επειδή δεν θέλουν αγαθοεργίε, ε, εκεί πρέπει να κοπεί η βοήθεια, το λέτε και το υποστηρίζετε επισήμω. Απάντηση. Η Save the Children θεωρεί ότι η βοήθεια πρέπει να πάει εκεί που τη χρειάζονται, σε αυτού που τη χρειάζονται περισσότερο από αυτού που έχουν μείνει πίσω, όπω τα παιδιά και το μίσα που τα επηρεάζουν άμεσα. Τώρα, κατά πόσον αυτό είναι συμβατό με την προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα. Είναι προφανές το ερώτημα και ρητορικό. Μήπως είναι λίγο πρόωρο το να αλλάξουμε το δίκτυο του Εκρεμούς αυτού και να περάσουμε από παραδοσιακούς τόπους χορήγησης βοήθειας στην υπόθεση πως ο ιδιωτικός τομέας είναι η πανάκια. Θα επανέλθουμε λίγο συντονιστής στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω όμως να μιλήσουν και οι υπόλοιποι του πάνελ Στι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, ε, να δούμε που ε, υπάρχουν εμπόλεμοι σειράξει. να βοηθήσουμε σίγουρα. Ε, σημαντικά είναι αυτά και όπως και ο Σάρλ θα πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη στην ηγετική θέση και να βοηθήσουμε τα δρόμια δικαιώματα. Συμφωνείτε? Διαφωνείτε? Σηκώστε τα χέρια άμα διαφωνείτε. Σκέφτεστε το Ιρλανδικό backstop, σηκώστε χέρια. Σε εσά κύριε θα έρθω μετά. Αλλά είναι σοβαρά αυτά τα θέματα. Πηρεάζει και το πολιτέ δημοσιονομικό. Νίσον. Νόρμπερτ Νόιζερ λέγομαι. Είμαι από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και θα τα πω γερμανικά για να κάνει και ένα διάλειμμα για καφέ η γερμανική καμπίνα. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση η οποία σχετίζεται με το θέμα ειρήνη, ασφάλεια, ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική που είναι έντονα προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, για να μην πω καταπολέμηση, και το λέω συνδυτά, καταπολέμηση της μετανάστευσης. Όλα τα βλέπουμε από αυτό το πρίσμα και εξού και λαμβάνονται διάφορα μέτρα ασφαλείας, ε, τα οποία συγχρηματοδοτούνται. Και παίρνουμε κονδύλια από τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για αυτό το σκοπό. Εγώ νομίζω ότι ως πολιτική που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της ανάπτυξης, θα πρέπει να πούμε ότι η αναπτυξιακή πολιτική πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την καταπολέμηση της φτώχειας φτώχεια. Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Και αν τώρα θέλουμε πρόσθετα μέτρα να υιοθετήσουμε για τη σταθεροποίηση, παραδείγματο χάρη ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών, αν θέλουμε στήριξη των στρατιωτικών αστυνομικών δυνάμεων, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αν αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, ναι, να χρηματοδοτηθεί, αλλά με άλλα κονδύλια. Όχι με κονδύλια τα οποία προβλέπονται για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Πολλές φορές ακούσετε από τις ομάδες προβληματισμού και τα think tank να λένε ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αν δαπανούμε χρήματα για να προσπαθήσουμε Τέλο πάντων, πώ να το πω, ότι μπορεί να ε, είναι τρόπο αντιμετώπιση μετανάστευση βοήθεια, δεν είναι σωστό. Γιατί είναι ανάλογα τα δύο μεγέθη. Όταν αυξάνεται το ένα, αυξάνεται και το άλλο. Δεν θέλω να σα αφήσω εκτό, αντεμπάγιο. Ε, πρώτα απ' όλα, εσεί να πάρετε το λόγο, γιατί συζητούμε διαμετρώντα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, τι ε, συγκρούσει και τι εμπόλεμε καταστάσει στην Αφρική. Το βλέμμα μα είναι στραμμένο πολλών στην Αφρική όταν συζητούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που βλέπουμε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Κοινά είναι τα προβλήματα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής ή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Αφρικής. Κοινά τα προβλήματα. Κάποιοι τα είπατε προβλήματα από των ανθρώπινο δικαιωμάτων. Άρα, ανεργία, φτώχεια, ανισότητες. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ είναι σημαντικό να αρχίσουμε κάπως να δομούμε την όλη συζήτηση με βάση όχι τόσο την υπόθεση ότι μια περιφέρεια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτό εγώ που λέω μονοπόλιο των λύσεων και μια άλλη περιοχή έχει το μονοπόλιο των προβλημάτων. Όχι, αν ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση, η συζήτησή μας ε, δεν θα βοηθήσει. Δεν θα ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την καινοτομία και μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό πειραματισμό, αλλά θα παίξουμε παιχνίδια ισχύω και σχεσμό δυνάμων. Μια κυρία είπε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ξαναγίνει μεγάλη. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε και εμένα με ενδιαφέρει και με ανησυχούν πρέπει να σας πω ορισμένες εξέλιξεις που έχουν να κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και των πολιτών σε ορισμένες από τις ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ε, να το δούμε αλλιώ. Πώς θα κάνουμε τον κόσμο μεγάλο ξανά, όχι την Ευρώπη μεγάλη ξανά. Αυτό είναι νομίζω το θέμα μας. Ε γιατί πρέπει να βάλουμε να συζητήσουν ε, ποιοι. Η Αιθιοπία, εκεί που ζω, και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Αν γίνει αυτό, ε, θα είναι όχι μονόπλευρο, που η μία πλευρά θα κάνει κηρύγματα στην άλλη, αλλά θα είναι αμοιβαίο ο όφελος μιας τέτοιας συζήτησης για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και αυτό έχει να κάνει με όλο το φάσμα των αναπτυξιακών θεμάτων. Θέλουμε να δώσουμε επίσης και πραγματικό νόημα στην ιδέα ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ανήκουν σε όλους μας. Δεν είναι απλά ένας ευγενικός τρόπος να μας κάνει κάποιος να νιώσουμε καλύτερα. Όχι, δεν αφορά μόνο την Αφρική, αφορά και τη Λατινική Αμερική, κάποια μέρη της Ασίας κτλ. Όχι, είναι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορούν τους πάντες. Και θα πρέπει να τους επιτύχει όλη η ανθρωπότητα. Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα γίνουν λειτουργικά. Ξέρουμε ότι η Αφρικανική Ένωση έστειλε μια αντιπροσωπεία και να ζητήσει, να ζητήσει να δικαιώματα αυτό λες. Ναι, ναι, Υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να γίνει αυτό. Έχουμε πρώτα-πρώτα τα δικαιώματα των μεταναστών. Όλα αυτά που γίνονται στην θάλασσα καταπατούν τελείως το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα. Η Δημοκρατική Αφρική ρωτάει, απευθύνεται στην Ένωση. Μα τι, τι στο διάλογο γίνεται σε διάφορα μέρη της ε, Ευρώπης. Στο Αμπιτζάν είδατε τι γίνεται. Στην συνάντηση κορυφής είπαν οι Αφρικανικές χώρες, θέλουμε αυτό να μπει στο τραπέζι. Μην θέλετε μόνο ένα πρόβλημα ε, ευρωπαϊκό. Να κάτσει να μα εξηγήσει ο ή άλλο. Θα ήθελε να έρθει εδώ με την προσωπή Αφρικανή Ένωση και να μιλήσει για το μεταναστευτικό στη Μεσόγειο. Σηκώστε τα χέρια. Σηκώστε τα χέρια, διαφωνείτε τώρα. Α, βλέπω ότι υπάρχει ευρύ υποστήριξη τη ε, ιδέα σα. Την τελευταία φορά που ήρθατε, μιλήσαμε για ε, σύγκρουση, για ανθρώπινα δικαιώματα και ακριβώς τα πλαίσια της Ευρώπης τα είχαμε πει τότε. Ναι. Άλμπεκτσεν. Προσοχή, προσοχή. Να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την αναπτυξιακή αρρωγή και τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, πρόκειται για θεματολόγιο μετασχηματισμό του κόσμου αλλά και της Ευρώπης. Οπότε είναι επικίνδυνο να μιλούμε για στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως να πρόκειται ε, για ένα σύνολο στόχων ανεκπλήρωτων. Μα θα έχει αλλάξει η όψη ε, του, του, του κόσμου σε λίγα χρόνια. Μα όλα αυτά είναι κατεπήγοντα. Όλα αυτά αφορούν κάποιο είδου αγανάκτηση, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τους στόχους ανάπτυξη. Ε, ανάπτυξης. 5, το 10, τι γίνεται με την ανισότητα τι γίνεται με τα ανισότητα όσον αφορά την ανεψυχική πολιτική της Ευρώπης. Μέσα στην Ένωση φουσκώνει το ποτάμι της ανισότητας. Ε, ασφάλεια και ανθρώπινα δικαιώματα. Για να το δούμε λίγο. Είναι πολύ επικίνδυνο να μπλέκουμε το, θέμα του στόχου 16 όσον αφορά τις συγκρούσεις. Και υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το πώς θα σταματήσει η αντιμορρησία κράτος δικαίου, προστασία ανηλίκων, προστασία γυναικών από τη βία που υφίστανται κάθε μέρα πέρσι. Δημοσιοποίησαμε μία έκθεση εδώ στις Βρυξέλλες. Ούτε μία γυναίκα στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να κυκλοφορεί το βράδυ αισθανόμενη φόβο. Γιατί όλα αυτά που λέμε για τιμωρησία, για ασφάλεια, προστασία από τη βία, όλα αυτά είναι κάτι καθολικό, παγκόσμιο. Άρα αυτό θέλω να ακούσω από εσά σήμερα εδώ. Τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά, τι θα γίνει να έχουμε κάποιο είδου ε, επεξεργασία φεμινιστικής πολιτικής και μέσα από την εξωτερική πολιτική, γιατί έχουμε ε, κορυφαία εξέχοντα μέλη που δεν, ε, που δεν κάνουν τίποτα ή απουσιάζει ο φεμινισμός από τα έγγραφα της Ένωσης, δηλαδή μια αναπτυξιακή πολιτική που να έχει ως αυθετηρία την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην κοινωνία, στις κοινωνίες και έτσι να γίνει ο μετασχηματισμός. Αυτό θα πρέπει να διαπνέει την πολιτική. Δεν είχαμε πει να μας το γίνει πιο συγκεκριμένη ανισότητα από Δευτέρα το πρωί. Ναι, μια φεμινιστική αναπτυξιακή πολιτική θέσεις απασχόλησης, για τις γυναίκες. Εγώ μιλάω για αυθεντικά φεμινιστική πολιτική. Λέω κύριε Άλμπριτ, χτσεν. Όχι, όχι, μιλάω για τη συρρήκνωση των θέσεων απασχόλησης, για προγράμματα, για χρηματοδότηση, τι μπορεί να κάνουν οι ΜΚΟ. Σάρλ, τι λες. Ναι, Σίγουρα ε, υπάρχουν και φτωχοί στι πλούσιε χώρε, υπάρχουν και φτωχοί χώρε μέσου εισοδήματο και υπάρχουν φτωχοί στι πολύ λίγο αναπτυγμένε χώρε. Και οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη μα υποχρεώνουν να δώσουμε μια απάντηση σε όλα τα προβλήματα, όπου και αν βρίσκονται οι φτωχοί στι λιγότερο αναπτυγμένε, στι μέσου εισοδήματο, στι ε, ανεπτυγμένε χώρε. Όλε οι χώρε που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις και συμφωνούν είναι ότι θα πρέπει ο καθένας να αναπτύξει τη δική του στρατηγική για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Αλλά θα πρέπει να έχουμε διάλογο ή θα απλώς θα περιοριζόμαστε να είμαστε οι πρώτοι δωρητές στην Αφρική ή ε, να πάρουμε στα σοβαρά τους στόχους τη βιώσιμης ανάπτυξης. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι σε κάθε χώρα σε επίπεδο εθνικό και στο κοινοβούλιο και στο, στην κυβέρνηση θα λαμβάνουμε τα μέτρα μας ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους. Συνδεμή θα έχουμε τις λατινοαμερικανικές εξέλιξεις στην Αφρική. Λίγους πλούσιους και πάρα πολλούς φτωχούς. Και στο Μαλαού υπάρχει μια ανακατανομία με τι άλλο. Και ακόμη και αν έχουν ελάχιστου πόρου, τουλάχιστον κάνουν μια καλή ανακατανομή γιατί έχουν ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, ένας έξυπνος τρόπος ανακατανομής ε, του εισοδήματος και μείωση των ανισοτήτων. Και ο ιδιωτικός κλάδος διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Πώς θα μπορούσαμε να τον αποκλείσουμε. Οι κυβερνώντες και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα εφαρμόσουν ε, στη χώρα τους. Όχι εμείς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να πούμε δεν θα σας αναπτύξουμε εμείς, εσείς θα αναπτυχθείτε, εμείς θα σας συμπαρασταθούμε έχουμε κάποια πείρα και μπορούμε να σας ε, βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων, γιατί και εμείς είχαμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ένα μοντέλο που θα μπορούσε να γίνει παράδειγμα προς ή να είναι πηγή έμπνευση και για άλλους. Επίσης, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την αρχή της διαφοροποίησης, γιατί αυτή η αρχή αποκλείει από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια τις χώρες μέσου εισοδήματο. Και θέλουμε να εξαλείψουμε την ακραία φτώχεια στον κόσμο, θα πρέπει να φροντίσουμε οι παν-φτωχοί, όπου και αν βρίσκονται ε, να βοηθηθούν. Και οι περισσότεροι βρίσκονται στι χώρε μεσαίου εισοδήματο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάλογο με αυτέ τι χώρε και να του πούμε είστε οι πρώτοι υπεύθυνοι. Και δεν θα σα δώσουμε χρήματα γιατί έχετε αρκετού ε, πόρου και έχετε αρκετό πλούτο. Αλλά εσεί θα πρέπει να υλοποιήσετε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εσείς πρέπει να αλλάξετε την πολιτική σας. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τεχνογνωσία, με τεχνική αρρωγή. Και αυτή θα πρέπει να είναι η μερίδα του μέλλοντος. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο αυτή η μερίδα του μέλλοντος επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά σε επίπεδο τεχνογνωσίας, μετάδοσης γνώσης, ε, ανταλλαγής εμπειριών, μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινωνικά μοντέλα, προβάλλοντας τα δικά μας κοινωνικά μοντέλα, την φοροληπτική μας ικανότητα, την αναδιανεμητική μας ικανότητα, να τους βοηθήσουμε να ενεργοποιηθούν και να αλλάξουν την πολιτική τους. Γιατί λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει επαρκή δέσμευση μερικές φορές των κυβερνήσεων ή τουλάχιστον με συνέπεια. Μακάρι αν θα μπορούσαμε να γράψουμε σε ένα φύλλο χαρτί πώς θα αναγνωρίζετε μια φεμινιστική αναπτυξιακή πολιτική, αν εμπρικείτε κι εσείς, ε, Σαλ. Γράψτε μου σε ένα φιλοχαρτί ε, το κατάλογο χωρών που επειδή είναι χαμηλ... μεσαίου εισοδήματος δεν δικαιούνται στο μέλλον επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Κάποια ζήτησε το λόγο κάπου στη μέση. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. και μετά θα δώσω το λόγο στην Άταλη. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μίρια Μπλάσολ. Είμαι πρέσβης της ε, Ουγγάντας στις χώρες Μπενελούξ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μία παρατήρηση σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία για το Save the Children και την Αφρική και το κατά πόσο ε, χρειάζεται ίδιο επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας η Αφρική. Στην Ουγκάντα είχαμε μια μακροχρόνια πολιτική όπου ζητήσαμε εμπόριο και προτιμούμε το εμπόριο από τη βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια ακόμη στην Ουγγάντα, αλλά το τμήμα της βοήθειας θα θέλαμε να ευνοεί το εμπόριο. Και νομίζω ότι περισσότερες αφρικανικές χώρες αυτό θέλουν, ε, ε, κυρίως ε, βελτίωση των υποδομών. Η Λίντα Μακάβαν μίλησε για την φεμινιστική σκοπιά Πρόσφατα, μια μη κυβερνητική οργάνωση έλαβε κονδύλια και μάλιστα πήρε και βραβείο για το ψηφιακό κόσμο και την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη. Αυτό που έκανε για τις, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ζήτησε να συμβάλλουν στην εταιρική να συμβάλλουν και να δώσουν σε ένα μικρό χωριό στην ε, Ουγγάντα σε 150 ανθρώπους ε, κινητό και ε, έδωσαν 30 ευρώ στο κάθε παιδί και μάλιστα το έδωσαν όχι στους επικεφαλής οικογένειας, στους άνδρες αλλά στις γυναίκες γιατί θεωρούσαν ότι θα έκαναν πιο υπεύθυνη χρήση αυτών των κονδυλίων. Τώρα, 60 ευρώ το μήνα κάθε, ε, για έναν ε, ενήλικα στην ε, Αφρική είναι τεράστιο ποσό. Και χάρη σε αυτή την ενίσχυση έχουμε περισσότερη, περισσότερα παιδιά στα σχολεία, καλύτερη πρόσβαση στην υγεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση και σε επιχειρηματικό επίπεδο στην αυτοπασχόληση στην Ουγκάντα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο παρέχετε την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό, αυτή θα ήταν η παρατήρησή μου. Ο Άντριξ Πίμπαξ θα συμφωνούσε μαζί σας. Ήταν κατά της ε, χρηματοδότησης υποδομών στην Αφρική και μάλιστα μείωσε τη χρηματοδότηση των υποδομών. Αν ακολουθήσουμε τη δική σας πρόταση και επικεντρωθούμε στην οικονομική ανάπτυξη, που είναι μια πολύ αξιοσέβαστη ε, άποψη, ίσως θα πρέπει να μειώσουμε και τα ειδικά κονδύλια που προβλέπονται για τον κοινωνικό τομέα. Γιατί σε τελική ανάλυση τι σημαίνει προγραμματισμό, σημαίνει επιλογή. Οπότε άλλη πρόκληση για τους ευρωβουλευτές και το πάνελ μας είναι ποια είναι η ισορροπία μεταξύ ε, των δαπανών στην ε, ανάπτυξη και των δαπανών στην οικονομία, στην οικονομική ανάπτυξη. Και μια και τελειώνουμε αυτό το θέμα τη ασφάλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ένοπλων σειράξεων, ίσω είναι ατέλει να προσθέσει κάτι. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι που ανέφερε η Τζάκη για τη βοήθεια και την φιλανθρωπία ε, για την Αφρική αλλά και για άλλες ε, χώρες και περιοχέ του κόσμου. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε εδώ το ε, θέμα του ενδιαφέροντος ή του συμφέροντος δεν το κάνουμε από αγαθοεργία, από φιλαθροφία, αλλά είναι προ το συμφέρον μα και το δικό μα και τη Αφρική. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρίσμα του συμφέροντο, έχουμε τελείω διαφορετική αντίληψη τη κατάσταση. Δεν μιλούμε μόνο για αναπτυξιακή συνεργασία, μιλούμε και για το εμπόριο. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο για το εμπόριο. Βοηθάμε και για τη μετανάστευση. Και επίση έχουμε και την ανθρωπιστική ενίσχυση, συνεργασία για την ασφάλεια Οπότε συγκεντρώνουμε τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούμε ε, και τα αξιοποιούμε όλα για να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης είπατε να μην επικεντρωθούμε μόνο στην εξάλληψη της φτώχειας. Εδώ διαφωνώ. Γιατί Ελπίζα να ήμουν σαφή στην αρχή και θα πρέπει να προσέξουμε να μην συρρυκνώσουμε υπερβολικά το θέμα της ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αφετηρία, αν είχαμε σημειώσει πρόοδο με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είμαστε ακόμη στη θεωρία, στην πράξη χωλένουμε. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξης και νομίζω ότι η σημαντικότερη πρόκληση είναι το είδος της πολιτικής που θα έχουμε. Κυρίως εδώ και στο Κοινοβούλιο. Τον επόμενο Μάιο αυτό το κοινοβούλιο ή το επόμενο κοινοβούλιο θα θέλει να επενδύσει γιατί το θεωρεί προς όφελός του, προς το συμφέρον του να επενδύσει σε χώρες που είναι μακρινές, που ξεπερνούν τα δικά του σύνορα. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση στο μέλλον. Νομίζω ότι υπάρχει μία ταραχώδης κατάσταση όταν μιλούμε για τη, τις σειράξεις, ε, τη σταθερότητα, την φτώχεια και το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Μετά την τελευταία έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες ε, από το πάνελ για το κλίμα, έχασα τον ύπνο μου, γιατί εκεί διάβασα ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να πετύχουμε το 1,5 λίγο παραπάνω ακόμη το στόχο των Παρισίων δηλαδή τη Συμφωνία των Παρισίων και μια και δεν είναι περιθωριακό πια το ζήτημα γιατί πριν από λίγα χρόνια είχαμε τη φατρία της ανάπτυξης και τη φατρία του περιβάλλοντος και σπάνια μιλούσαν μεταξύ τους. Τώρα και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να τα ενοποιήσουμε όλα αυτά και μάλιστα να δράσουμε και άμεσα Έχω τρεις ιδέες να προτείνω. Η Γαλλία πρόσφατα εγκαινίασε τη νέα της αναπτυξιακή πολιτική και ένα από τα στοιχεία της πολιτικής αυτής είναι η ιδέα 100% Παρίσι, δηλαδή ε, συνεκτίμηση του κλίματος ε, σε ο, στο σύνολο του αναπτυξιακού προϋπολογισμού. Και με τη κυβέρνηση Ομπάμα είχαμε κάτι αντίστοιχο. Είναι απολύτως απαραίτητο λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, ε, αφιερώσει την κλιματική πολιτική το 25% μόνο του προπολογισμού, αλλά να έχει να συνεκτιμά τις κλιματικές αλλαγές σε όλες τις πολιτικές. Δεν σημαίνει ότι όλα τα, όλα τα χρήματα θα πάνε στο κλίμα, αλλά οι δαπάνες να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξοδεύει 112 δισεκατομμύρια το χρόνο, το χρόνο όχι ανά 7 αιτία, σε επιδοτήσεις για τα ορεκτά καύσιμα, ενώ υποσχέθηκαν ότι μέχρι το 2020 θα τις καταργήσουν. Το θέμα είναι όχι ότι ενισχύουν μόνο το πρόβλημα, αλλά ότι αφαιρούν επενδύσεις από το τρίτο σημείο, που είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πιο άμεσα στις μεταβάσεις, στην ενεργειακή μετάβαση, στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στη μετάβαση στη γεωργία, στη διαχείριση του ύδατος. Αυτά είναι όλα απολύτως απαραίτητα για να ανατρέψουμε τις τάσεις. Αυτές είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες, κατά τη γνώμη μου, για να μειώσουμε τη φτώχεια και να λάβουμε υπόψη και το κλίμα, γιατί είναι αλληλένδετη στόχη με οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε τώρα το πρόβλημα, σε 10 χρόνια θα έχουμε τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αν δεν λάβουμε μέτρα τώρα. Κάποιο εκεί πίσω ήθελε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ Σάιμον. Άντολφ Κλούκελε, λέγομαι από το Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υπό ε, την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Εθνών. Ο τίτλος είναι «Καινοτομία και Ανάπτυξη». Και αυτό που βλέπω κάποιοι, τουλάχιστον συζήτηση, να οπισθοχωρούν σε παραδοσιακά μοτίβα συζήτησης, αυτά που βλέπαμε πριν 15-20 χρόνια. Η Άννα Μπίργκιτ νομίζω τα είπε πολύ καλά για την, τον καινοφανή χαρακτήρα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό που μου λείπει από αυτή τη συζήτηση, εν μέρη προέκυψε στην τελευταία παρέμβαση. Αφενός θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα ε, που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετατοπίζονται σε άλλες χώρες, κλίμα κτλ. Αλλά επίσης πώς μπορεί να μας καθοδηγήσει αυτό, αυτή η δέσμη στόχων στις σχέσεις μας με η Ρωσία, Κίνα, κτλ. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε το θεματολόγιο μόνο σε ένα ε, μέρος χωρών με μεσαίου εισοδήματος, για παράδειγμα. Είναι μικρό αυτό το κομμάτι χωρών. Hello, um, I'm... Γεια σας. James Ingram. Μια οργάνωση διεθνής για προστασία της φύσης για την αλλαγή του κλίματος. Ε, θα έλεγα ότι δεν είχε αναφερθεί, ευτυχώς με πρόλαβε κάποιος. Φαντάζομαι ότι είδατε αυτό το γράφημα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τη βιοσφαίρα και το τι γίνεται. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη βιοσφαίρα, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να ιεραρχήσουν προτεραιότητε. σω εκεί θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη μέγιστη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα ζητήματα αυτά τη βιοσφαίρας κατά προτεραιότητα. Να βγάλουμε τον κόσμο από τη φτώχεια με αυτόν τον τρόπο και να βοηθήσουμε και το περιβάλλον. Εκεί εστιάζουμε κατά την άποψή μου και θα πρέπει να εστιάζουμε. Στο Αφγανιστάν φέτος από την ξηρασία παρά τους Ταλιμπάν εκτοπίστηκαν περισσότεροι. Και τα πράγματα θα επιδεινωθούν και αν δεν ε, το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, πράγματα που μας φαίνονται σήμερα μικροπροβλήματα θα επιδεινωθούν, θα διωγγωθούν στο μέλλον. Κάποιος άλλος θα θέλει να λάβει το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, πέντε λεπτά θα εστιάσουμε στην παγκοσμιοποίηση. Θα ζητήσω μετά από του ε, πανελίστε να συνοψίσουν και να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα, ώστε μετά να δώσουμε τη σκητάλη στη Φεντερίκα Μογκερίνη και τον Bill Gates. Αυτή είναι η τελευταία σα ευκαιρία λοιπόν να συνεισφέρετε στα ζητήματα που έπρεπε να κάνουμε την ανάπτυξη, το εμπόριο, την παγκοσμιοποίηση, την ανάπτυξη. Παρακαλώ. Γεια σα. Είμαι ασκούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να συνεχίσω ε, από εκεί που σταμάτησε ο προελαλή σα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα μπορούσε να της μεγαλύτερη ισχύ στο μέτωπο των διεθνών σχέσεων. Ε, ξηρασία, είπε ο πρόεδρος σας. Γενικά, κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε συγκρούσεις και πολέμους, όπως στη Σύρια, για παράδειγμα. Ε, που παρότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Απ' την άλλη έχουμε την Ιεμένη, τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα, ανθρωπιστική καταστροφή. Δεν δίνεται όμως ε, ιδιαίτερη έμφαση ούτε ενέργεια επαρκής ε, δαπανάται για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Άρα και αυτό να το λάβουμε υπόψη στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. David θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Αφρικής. Και είναι και πιο νέος ο πληθυσμός, ενώ γυράσει και ε, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ε, με όλα αυτά τα επιβαρυντικά για τα συνταξιδοτικά στήματα, στη μετάσφαση κτλ. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκροτήθηκε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για να συζητήσουμε τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής με τρεις ηγέτες κρατών, τέος ηγέτες κρατών από αφρικανικά κράτη. Κανείς δεν ζήτησε χρήματα Απλά ζήτησαν αλλαγή ε, στους συσχετισμούς ε, ισχύω και εξουσία. Να μπορούν δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Δέλτα Τάφνα, να εκπροσωπούνται οι Αφρικανοί περισσότερο ή στο ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Και για το πολιτισμικό πλαίσιο, 140 δις ευρώ θα πρέπει να διατεθούν στην καταπολέμηση της φτώχειας. Με στόχο τους κοινωνικούς τομείς και τις πιο φτωχές χώρες. Όμως υπάρχουν και άλλα θεμελιώδη ζητήματα, διακυβέρνηση, χρηματοπιστωτικό απόρριτο κτλ. Εμπόριο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτά, αλλιώ δεν θα μπούμε στην ουσία και δεν θα έχουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Inequality Παγκοσμιοποίηση και ανισότητα συνδέονται άρρηκτα. Στη δική μου χώρα Έχουμε πάρα πολλέ αιτίε που υπάρχουν οι ανισότητε. Τους καλομαθημένους, τους υψηλόμιστους και που αναφερθεί είναι η αποβιομηχάνηση και βλέπουμε για αυτό το λόγο ότι στην Κίνα είναι δύσκολο να ε, βρεθούν κάποιες λύσεις. Επομένως, Υπάρχουν από την ανισότητα από κάτω οικονομικοί παράγοντες. Παλεύουμε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν η Λίντα θέλει να πει κάτι πριν επανέλθω με το πάνελ στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουμε τους παγκόσμιους μοχλούς ε, και παράγοντες ανισότητας. Ίσως θα μπορούσε να μας δώσει την εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι από αυτούς τους μοχλούς παράγοντες ανισότητας στα δικά μας κράτη-μέλη. Είναι αυτοί που καθορίζουν και το θετικό πλαίσιο το οποίο εμείς προσπαθούμε να καθορίσουμε, πιέσει μεταναστευτής και τα λοιπά. Έχουμε λαϊκιστικά κόμματα. Κάποιος ρώτησε πώς θα είναι το Μάη το νέο κοινοβούλιο, το Μάιο του 19. Ίσως ε, δούμε λαϊκιστικά κόμματα και τελείω διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις εδώ. Όχι μόνο στην Κοινοβουλία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα κράτη-μέλη ορίζουν ε, του επιτρόπου και μπορεί να είναι τελείω διαφορετικέ πολιτικέ. Ακούσαμε κάποιες κριτικές για κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Αυτά θα στείλουν επιτρόπους εδώ για την επόμενη θητεία. Είναι πάρα πολύ διαφορετική συζήτηση, Σάιμον. Λες, ναι, να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το Brexit πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από ανθρώπους που ένιωθαν ότι τους είχαν αφήσει πίσω. Ε, για κάποιον ε, εκλογική μου περιφέρεια, το πρόβλημα ήταν το σύστημα ασφάλισης, ότι δεν είχαν δουλειές στην Βορραλία κτλ. Πώς αυτό επηρέασε τώρα την αυξιακή πολιτική. Και έχουμε αυτό το πολιτικό πλαίσιο. Σε αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούν οι πολιτικοί. Μα έτσι αποφεύγουμε την ουσία επί της οποίας πρέπει να νομοθετήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Να είπατε για την ασφάλεια, είπαμε, ε, πρέπει να δαπανίσουμε για αυτά, για το μεταναστευτικό. Ε, ο Νόρμπερτ είχε πάει σε κάποια συνάντηση, αναφέρθηκε ο στόχος 16, αλλά είπαμε ότι αν δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν μπορεί να υπάρξουν και επενδύσεις, δεν μπορεί να κατευθούν και κονδύλια. με τον προπολισμό, χωρί τον προπολισμό, τι να κάνουμε. Έτσι θα πρέπει να προσαρμοστεί η χρηματοδότηση τη Ένωση. Δεν είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι έχουμε αυτό τον κουμπαρά για την ανάπτυξη και χωριστά να βγάλουμε λεφτά για την ασφάλεια. Μα δεν θα το δείχνουν τα κράτη-μέλη. Δεν θα εγκριθούν τόσο πολλά λεφτά. Άρα μην αποφεύγουμε να συζητήσουμε για αυτά που πρέπει να νομοθετήσουν οι πολιτικοί. Θα πρέπει στην Ελλάδα να δώσουν τη μάχη τους στις εκλογές, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στους ψηφοφόρους. ο κόσμο μπορεί να το αποδεχτεί ότι πρέπει να συνεργαστούμε με άλλε χώρε για το μεταναστευτικό, αλλά θέλουν αποτελέσματα και είναι δύσκολο ε, Εμεί οι πρωτευτικοί αριστεροί να βρούμε απλέ ε, ε, Δεν είναι δυνατόν να βρούμε τι εύληπτε λύσει συνένεση εδώ, συνένεση στο Συμβούλιο και έτσι να προωθηθούν οι πολιτικές που περισσότερο θέλουμε να δούμε. Άρα χρειάζεται βαθύτερος προβληματισμός γι' αυτά. Να σας πω τι έγινε εκεί που κλείσαν τα ανθρακοριχεία. Τι έγινε με τη διάλυση του κοινωνικού ιστού και που καταλήξαμε μετά από όλη αυτή τη διαδρομή στο λαϊκισμό του Brexit. Έχουμε, έχουμε λίγη ώρα μέχρι να έρθουν οι προσκεκλημένοι μας και τώρα ξεκινούμε με την Νατάλη και καταλήξουμε στον Σάρλ στην άλλη μεριά. Τα ερωτήματα ήταν τι θα πρέπει να γίνει με τρόπο διαφορετικό και άλλο ερώτημα ήταν τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, θα πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη. Μα στις Βρυξέλλες εύκολα κανείς γλιστράει σε κάποια τεχνοκρατική συζήτηση για το πολίτες πλαίσιο. Θα πρέπει να διατίθενται κονδύλια, θα πρέπει να γίνει με τον α ή β τρόπο, μα όλα αυτά όμως είναι δευτερεύοντα. Τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξη είναι αυτά που ε, σήμερα συζητούμε. Φεμινιστική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, βοήθεια ε, αλλά μην το παρακάνουμε. Τι γίνεται με τις άλλες προκλήσεις, τη μαγκοσμιοποίηση και σε έξι μήνες έχουμε εκλογές. Μα για την ανάπτυξη χρειάζεται κάθε κόμμα να έχει ένα μανιφέστο και όλοι μαζί να κερδίσουμε την μάχη της ανάπτυξης για την επόμενη εξάμεινο. Πέστε μας, πώς θα τα καταφέρουμε. Τέσσερα πολύ σύντομα σχόλια. Ένα εξαιρετικά συνοπτικό γιατί ήδη το είπα. Όχι υπερβολική συρρήκνωση ή μείωση. Και φυσικά να αξιοποιήσουμε τη μέχρι τώρα πρόοδο και να την διευρύνουμε. Δεύτερον, ακριβώς λόγω της ανάγκης χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και όχι απλώς μεταφορά των κονδυλίων. Και τρίτον, Περάστε από τα λόγια στα έργα. Αφήστε τα λόγια μόνο για την κοινή προσέγγιση. Όταν μιλούμε για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, για διοργανική συνεργασία, για διακλαδική συνεργασία, γιατί είχαμε κάποια επιτυχία, ίσως μεγάλη μεταξύ της ασφάλειας και της ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και την ανθρωπιστική πτυχή και την περιβαλλοντική, και ούτω καθεξής. Και τέταρτο και πιο σημαντικό, ένα θέμα που σχεδόν δεν ε, αναφέραμε, είναι η πολυμέρεια. Ίσως ο Σάιμον το υπενήχθηκε. Αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να δράσουμε μόνο. Εμείς ως Ευρωπαίοι ίσως είμαστε οι μόνοι ή οι ισχυρότεροι ας πούμε που έχουμε απομείνει υπέρμαχοι της πολυμέρειας. Θα πρέπει όμως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο υπερασπιζόμαστε την πολυμέρεια. Γιατί για πολύ καιρό υπερασπιζόμασταν την πολυμέρεια συνεργαζόμενοι με τους ομοειδεάτες μας, χώρες ή ε, εταίρους. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι ομοειδεάτες, γιατί τώρα αλλάζουν. Δεν είναι πια η ίδια ομάδα. Για τους συγκεκριμένους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης έχουμε μία ομάδα μια συγκεκριμένη συμμαχία και ίσως κάποιοι παλιοί μας φίλοι γίνουν σημερινοί μελλοντικοί αντίπαλοι. Και όντως σε μερικά θέματα στόχων βιώσιμης ανάπτυξη είναι αντίπαλοι. Μας έχουν μείνει 11-12 λεπτά, 2 λεπτό καθένας λοιπόν από το υπόλοιπο πάνελ. Τρία σύντομα σχόλια. πρώτο να κάνουμε ό,τι είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να αποδείξουμε στον κόσμο ότι τα κονδύλια πιάνουν τόπο και να, δείξουμε, να αποδείξουμε στους εταίρους μας ότι οι επενδύσεις τους είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. Γνωρίζουμε από τις στατιστικές ότι η παγκόσμια μείωση της φτώχειας μπορεί να είναι, να είναι εφικτή. Και μπορούμε να επενδύσουμε χρήματα για να αποτρέψουμε τη μετανάστευση, να δώσουμε κίνητρα για τη μετανάστευση. Επίσης, να αναλάβουμε, να γιατί τι νόημα έχουν οι προτεραιότητες αν δεν υπάρχει ιεράρχηση. Θα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Χρειάζεται παγκόσμια μετάβαση από τη βρώμικη στην καθαρή ενέργεια. Αυτό θα μπορούσε να είναι το δώρο της Ευρώπης προς τις επερχόμενες γενναίες, αλλά θα πρέπει να ρεψοκινδυνεύσετε και να επενδύσετε τις επενδύσεις σας. Αν κάνετε κατακαιρματισμένη δαπάνη, θα έχετε πολύ περιορισμένη επιτυχία και ανεπαρκή. Και αυτό που ακούσαμε περισσότερο από αυτή τη συζήτηση είναι να εμείνουμε στις αξίες ε, και να τις υποστηρίξουμε. Οι αξίες που έκαναν την Ευρώπη δυνατή, που έκαναν τις ΗΠΑ δυνατές και τους έδωσαν ηγετικό ρόλο στον κόσμο, από αυτές τις ε, αξίες δεν πρέπει να υπαναχωρήσετε, γιατί αν υπαναχωρήσετε σε σχέση με τις θεμελιώδεις αξίες, όχι μόνο θα απογοητεύσετε τους ε, συμμάχους σας, και αυτούς που θέλουμε να υποστηρίξουμε, αλλά ουσιαστικά θα προδώσουμε τους εαυτούς μας. Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε και να δούμε ποιους θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Γιατί η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης είναι το θεματολόγιο του ανθρωπισμού. Να μπει ο άνθρωπο στο επίκεντρο του προγράμματος, Να δούμε και να επικεντρωθούμε στο τι λειτουργεί. Έχουμε μια πεντηκονταετία αναπτυξιακή συνεργασία και ξέρουμε ότι αν επενδύσουμε στι γυναίκε και τα κορίτσια θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Και επίση για την πολυμέρεια, να δώσουμε ένα βραβείο στην πολυμέρεια, να δημιουργήσουμε χώρο για εταιρικές σχέσεις και συνεργασία. Γιατί μιλούμε κυρίως ε, για τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα, αλλά δεν δίνουμε αρκετή τη φωνή στην κοινωνία των πολιτών. Γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερο κύμα πολιτών που απομακρύνονται, αποστασιοποιούνται και αρχίζουν και διαφορούν. Θα πρέπει αυτή την κοινωνία των πολιτών να τη φέρετε στις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ κάτι. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην αστίαση σε προτεραιότητες που καθορίζονται από τους εταίρους μας, αντί να προτείνουμε αντιπροτεραιότητες. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τοπικές προτεραιότητες. Γιατί δεν έχει νόημα να βάζουμε προτεραιότητες εμείς, να επιβάλλουμε τις προτεραιότητες σε άλλους, να ακούσουμε ποιες είναι οι δικές τους προτεραιότητες. <coughs> Ίσως σε αυτό δεν δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη δώσαμε αρκετή προσοχή σε κάποια είδη μακροοικονομικής πολιτικής που είναι σημαντικές. Και να επικεντρωθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο ότι γνωρίζουμε τι είδου οικονομικές πολιτικές λειτουργούν και τι, χρειαζόμαστε, τι οικονομικά χρειαζόμαστε στον κόσμο. Αλλά λυπάμαι, ένα σημαντικό τμήμα τη φτώχειας που δημιουργήθηκε ήταν το αποτέλεσμα της υπερβολική λιτότητας και μερικές φορές ήταν τελείως ανευνοήματος. Ε, ε, ενώ άλλες χώρες έχουν αποθεματικά δολαρίων στην Αφρική, ενώ σε τελική ανάλυση δεν επενδύονται αυτά στις υποδομές, ούτε επενδύονται στην παιδεία, ούτε στην επιστηστική ασφάλεια. Και παρόλα αυτά υπάρχουν οι πόροι για να γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω πού πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια, τα απορροφώνται από τη διαφθορά. Αλλά μερικές φορές είναι η μακροοικονομική προσέγγιση λάθος που αντί να υιοθετούμε μια αναπτυξιακή σκοπιά, υιοθετούμε τους δείκτες ε, της ε, μακροοικονομικής ε, προσέγγισης μόνο. Ο Σαργκέρες. Έχω τέσσερα σχόλια εδώ. Mm, Καταρχήν, οι ευρωεκλογέ θα λάβουν χώρα σε ένα πλαίσιο που, χαρακτηρίζεται από δύο κατηγορίες κομμάτων. Η μία κατηγορία κομμάτων ψάχνει μονίμως προβλήματα και η άλλη κατηγορία κομμάτων αναζητεί λύσεις. Αυτοί που αναζητούν λύσεις υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη πρόπτικη και δεν προβάλλεται αρκετά αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική. Θα πρέπει να βρούμε τα επιχειρήματα ε, για να να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τον κόσμο και να καταλάβει τι ενέργειέ μα. Δεύτερον, η Ευρώπη θα πρέπει να τηρήσει τι υποσχέσει τη, τι δεσμεύσει τη. Δεν αρκεί να έχουμε συγκεκριμένο ποσοστό επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να το τηρήσουμε γιατί 40 χρόνια ε, υποσχόμαστε αλλά και ανανεώνουμε τι υποσχέσει μα, αλλά δεν τι τηρούμε. Επίση, οι ε, στίχη βιώσιμη ανάπτυξη είναι καταθυντήρε γραμμέ. Δεν χρειάζεται να τα ψυρίζουμε. Οι στόχοι υπάρχουν, θα πρέπει να υλοποιηθούν και κάθε χώρα να έχει τη στρατηγική της για να τους εφαρμόσει. Ξεκινώντας από την Ευρώπη. Ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη έχουν στρατηγική για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ μία δεκαετία έχει μείνει για να τους υλοποιήσουμε. Θα πρέπει εκεί να είμαστε άψογοι ε, και άμεπτοι. Κάποιος είπε ότι δεν μιλήσαμε για την πολυμέρεια. Η μία της πολυμέρειας είναι τόσο σημαντική που το ανέφερα και στα εισαγωγικά μου σχόλια. Η Ευρώπη στο ισχύον πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την καταγγελία των είπα όλων των πολυμερών συμφωνιών, εμείς θα πρέπει να βρεθούμε στον προμαχώνα της υπεράσπισης της πολυμέρειας. Όσοι ενδιαφέρονται για μια πολιτική που θα στηρίζεται στο κράτος δικαίου και όχι στην ισχύ, ε, στη, στη δύναμη της πυγμής, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Επίσης προέκυψε από όλα τα σχόλια και τη συζήτηση ότι και στα θέματα συνέπειας πολιτικών έχουμε πρόοδο να σημειώσουμε. Θα σας δώσω μια, ένα παράδειγμα ασυνέπεια στην πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την έκθεσή μου για τη συνέπεια των πολιτικών και είχα προτείνει ε, να προβλέψουμε μια διαιτησία σε περίπτωση δύο, που δύο Υπουργεία ή δύο Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμφωνούν. Ε, σε τέτοια περίπτωση ο πρόεδρος αποφασίζει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο Πρωθυπουργό. Αλλιώς γίνονται άκαρπες ε, διπηρεσιακές ε, συνεδριάσεις ή σε διακυβερνητικό επίπεδο πάλι άκαρπες συναντήσεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και κατηγορηματικοί να προβλέψουμε ξεκάθαρους κανόνες. Και ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Μπορεί να είμαστε σκεπτικιστές, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε δραστήριοι. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και η Λίντα θα απαντήσει μετά με τις εικόνες, ε, τις φωτογραφίες με Γκερίνη και Bill Gates. Λοιπόν, το ETTG ενώνει 350 ερευνητέ από πέντε χώρες. Ε, θέλουμε να σκεφτούμε διαφορετικά την αναπτυξιακή συνεργασία, παγκοσμιοποίηση, ανισότητες. Θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά, όπως επίσης και την έλλειψη αηφορίας, ε, τις συγκρούσεις. Όλα αυτά τα θέματα συζητήθηκαν με τον τον άλλο τρόπο. Έχουμε ε, τις εκλογές, ε, έχουμε το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε τεχνικές προσαρμογές, κατά την άποψή μου. Πρέπει να ξεκινήσουμε ε, με τη βαθιά κατανόηση του πώς αλλάζει το θεματολόγιο. Έχω δύο ερωτήσεις Σηκώστε το χέρι αν συμφωνείτε με την πρόταση ότι πρέπει να γίνει συζήτηση για τη διεθνή ανάπτυξη τους μήνες που οδηγούν στις ευρωεκλογέ. Δεν συμφωνείτε, σηκώστε τα χέρια. Ωραία. Κάτι μετράει η συζήτηση. Κάπου οδήγησε. Και το τελευταίο. Το ETTG και η Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη ε, συνεργάζονται πολύ καλά. Θέλουμε να συνεχίσουμε. Αλλά το τελευταίο ερώτημα. Θα Έρθετε μαζί μας σε αυτήν την προσπάθεια. Σηκώστε χέρια. Εντάξει, τους υπόλοιπους δεν σας ρωτάω, μου φτάνουν αυτοί που σηκώσαν το χέρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αυτήν ε, την αίθουσα για τη συζήτηση που φυσικά και δεν κάλυψε τα πάντα. Πάρα πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς εδώ από το εξαιρετικό πάνελ. Our guest should be here within the next uh, seven minutes. Τα επόμενα 7 λεπτά θα είναι εδώ η προσκεκλημένα μας. Ε, αν θέλετε να τεντωθείτε, ε, έχετε 7 λεπτά. 4 ώρα θα ξαναξεκινήσουμε. εδώ μιλάμε κανονικά, ε. Τώρα ξέρεις, ε. then we then we go on a bit. Uh, just to let you know that that uh, Federica Mogherini and Bill Gates are running. Αργούν λίγο η Φεντερίκα Μογκερίνη και ο Μπιλ Γκέιτς. Ελπίζω όμως να μην ξεπεράσουμε την επίσημη ώρα λήξης της συνέντευξης. Σε πέντε λεπτά θα είναι εδώ, ελπίζω.

Um, good afternoon again everybody. Καλησπέρα σε όλους και πάλι σε αυτή την κατάμεστη αίθουσα. Έλεγα στον κύριο Γκέτς και κυρία Μογκερίνη ότι σπάνια είναι τόσο γεμάτε αίθουσε που βέβαια δείχνει το τεράστιο ενδιαφέρον για την σημερινή εκδήλωση. Καλώ όρισε ο κύριος Γκέτς, Ευρωβουλίο και καλώ όρισατε και πάλι Φεντερικά Μογκερίνη. Σήμερα θα συζητάσουμε το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής. Ήρθατε την πιο κατάλληλη ώρα. Έχουμε τέσσερις ευρωβουλευτές, νομοθέτες και σε συνεργασία με τους υπουργούς του επόμενους μήνες θα νομοθετήσουν, θα επεξεργαστούν μια πρόταση για ένα νέο πλαίσιο για την αναπτυξιακή μας πολιτική. Το σχέδιο της πρότασης το επεξεργάστηκε η κυρία Μουγκερίνη και το υπέβαλε και θα συζητήσουμε για τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και περιμένουμε ανυπόμονα να ακούσουμε όσα έχετε να μας πείτε. Ο Σάιμον Μάξουελ, εξ αριστερών μου, ο οποίος θα διευθύνει τη συζήτηση. Σάιμον. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή που ε, οργάνωσε την σημερινή εκδήλωση με μεγάλη μας ε, ικανοποίηση. Έχουμε αυτούς τους τρεις διάσημους προσκεκλημένους, την Φεντερικά Μογκερίνη, η πατή εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Bill Gates. Πού είναι ο Bill Gates? Και ο Ήμερ Σόλτ οποίο είναι επικεφαλή του Γερμανικού Αναπτυξιακού ιδρύματο. Είχαμε πάνελ, συζητήσαμε πριν, έρθετε εσείς και φτάσαμε στα συμπεράσματα ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι έχουμε σε 6-7 μήνες ευρωεκλογέ, θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να επερασπιστούμε την υπόθεση ανάπτυξη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντίρροπες δυνάμεις που θέλουν να δυναμητήσουν αυτή την ε, τάση, την ορμή που έχουμε τώρα. Επίσης θα πρέπει και να προβληματιστούμε όσον αφορά την ανάπτυξη σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, οπότε θα έχουμε όλο ένα και λιγότερες φτωχές χώρες γιατί ε, εκεί ζουν οι φτωχοί ε, μέσα σε χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις όπως αλλαγή του κλίματος. Τα συζητήσαμε όλα αυτά, ποιοι είναι χαμημένοι και κερδισμένοι τη παγκοσμιοποίηση και πώς θα έχουμε τελικά τον επιθυμητό μετασχηματισμό, τι θα γίνει το μεταναστευτικό, τις συγκρούσεις. Νέα, νέα θέματα στην υπόθεση ανάπτυξη. Και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της ανάπτυξης σε τεχνοκρατικό επίπεδο για τα χρηματοδοτικά μέσα, τη, τη, διαχείριση του προϋπολογισμού. Τέλος πάντων, ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Υπέρ της ανάπτυξης έχουμε τις δεξαμενές σκέψεις, πάρα πολλούς εκατοντάδες ερευνητέ και ιδρύματα υπό την σκέπη μας στο ETTG. Φαντέργα γίνει και Bill Gates. Θα μας μιλήσετε κι εσείς και είμαι... Κάντε τις εγγύσεις πριν τον Ήμερ. Και στο τέλος της συνάντησης, όταν θα έχετε φύγει, θα έχουμε τρεις, τον James Μάγκη από το ECDPM, του σε Σεμάστιν Τρέια, από το Παρίσι και το Φράγκα Έγγελ που είναι ένας από τους εισηγητές που θα μας μιλήσουν. Τότε, μετά. Φιντέρικα, ευθύς αμέσως έχεις τον λόγο. Να σας τα πω, να σε ικανοποιήσω, να σε ψυχαγωγήσω, με αυτό θα ήταν πρωτότυπο τέλος πάντων. Ποτέ δεν έχω δει στο κοινοβούλιο αίθουσα ή αδίποτε αίθουσα τόσο γεμάτη, ρεκόρ. Μακάρι να είχα τόσο κόσμο και στο Στασβούργο, όταν σας μιλάω στην Ολομέλεια. Τέλος πάντων, πολύ πολύ θετικό το ότι είσαστε τόσοι εδώ και από το Κοινοβούλιο και εκτό αυτού. Αυτό λέει πολλά για την διάθεσή σας, για τον προσανατολισμό σας, για το ότι θέλετε να συνεχίσουμε το έργο μας. Αυτά για αφετηρία, όχι, δεν ψυχαγωγεί αυτό, αλλά έτσι θυμόμαστε τις προτεραιότητές μας. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να έρθω σε αυτή την καταμεστή αίθουσα, στην αίθουσα Αλτσίντε Ντεγκάσπερη που με τιμά ιδιαίτερα και μιλούμε για την σχέση αναπτυξιακής εργασίας και καινοτομίας. Αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη. Για να αρχίσουμε με κάποια αριθμητικά στοιχεία. Για άλλη μια φορά, πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη επένδυσαν περισσότερα σαν αντοχική βοήθεια από όσο όλος μαζί ο υπόλοιπο πλανήτης. Πάνω του 50% της ε, αρρωγής προέρχεται από την Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει 20 δις ετησίως μόνο στην Αφρική. Αυτά δεν είναι δάνεια, είναι χορηγίες, είναι δωρεές για τις επόμενες γενναίες. Οπότε θα πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της προσπαθίας μας προς αυτή την κατεύθυνση και ξέρουμε ότι αυτά τα κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι για το δικό μας συμφέρον, ότι δεν είναι λεφτά πεταμένα. Ούτε νομίζω ότι κανένας πιστεύει κάτι τέτοιο. Ούτε καν φιλανθρωπία δεν το θεωρούμε. Δεν το κάνουμε αυτό επειδή είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι. Νομίζουμε ότι είναι μια έξυπνη επένδυση για ασφάλεια, σταθερότητα, ανάπτυξη. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, προκλήσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε την ιδέα της αντεξιακής βοήθειας, να γίνει πιο αποτελεσματική. Αλλάζει γρήγορα ο κόσμος και εντυπωσιακά. Και άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το πράγμα τον ίδιο τρόπο. Να τα κάνουμε, αλλά έχουμε την ευθύνη να σκεφτούμε το αύριο. Οπότε διερευνήσαμε νέους τρόπους αντισιακής συνεργασίας, ε, στη συνέχεια ε, του προσανατολισμού των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό, αυτό είναι ο μπούσουλας στην πολιτική μας αυτή. Η αφετηρία μας είναι η αλλαγή της μεθοδολογίας μας ως ένωση. Συνήθως κουράμε το δαχτώ στους άλλους, αλλά τώρα στραφήκαμε προς τα μέσα. Να δούμε εμείς τι κάνουμε και έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε το θέμα του 2030, διαμορφώθηκε μια συνένεση θεσμικών οργάνων, κρατών μελών, συντονισμός και αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά όσοι ξέρουν τα θεσμικά της Ένωσης ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πάλι όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία, δώσαμε περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο και οι επιπτώσεις των όσων κάνουμε είναι χωρίς προηγούμενο και άρα θα πρέπει συντονισμένα προς την διακατεύθυνση να πάμε έχω, έχω με αυτό, την, τον κοινό προγραμματισμό για όλο τον κόσμο και να κινητοποιήσουμε και άλλους όπως προτιμήσεις εμπορικές και συνεργασία ασφάλειας. Όλα αυτά, ό,τι έχουμε, ό,τι μέσα έχουμε, να τα συντονίσουμε. αυτό θα αλλάξει τα πράγματα. Άρα να αλλάξουμε το τι κάνουμε μέσα στην Ένωση και να αλλάξουμε και το τι κάνουμε με τους εταίρους μας. Πρώτα-πρώτα, συνεργασία με τον ΟΗΕ. Επίσης να συνεργαστούμε και με άλλους ε, οργανισμούς περισσότερο από ό,τι πριν. Τερίτων, προτεραιότητες με τους ε, κατατόπους εταίρους. Προσπαθούμε επομένως να βγούμε από την παραδοσιακή προσέγγιση δωρητή, δωρεοδόχο και να έχουμε αυθεντικές εταιρικέ σχέσεις, να αφουγκραζόμαστε πριν ενεργήσουμε και τέλος. Νέα μέθοδο συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σημαντικό. Πρώτα-πρώτα, εταιρική σχέση με τον ΟΗΕ. Ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουμε την πολυμέρεια που όπως σας είπα είναι ο μπούσουλα που έχουμε, είναι το να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και η Γενική Συνέλευση πριν από λίγε εβδομάδες συμφώνησε να εξυγχρονιστούμε στην συνεργασία μα για την ανάπτυξη, να αλλάξουμε τη μεθοδολογία μα για παντού στον κόσμο και να εξασφαλίσουμε ότι όταν αρχίσει να τρέχει ένα πρόγραμμα ποτέ να μην κάνουμε ό,τι γινόταν πριν από άλλους όπως από κάποιες φορείς του ΟΗΕ αλλά να αναβαθμίσουμε τι κάνουμε και αυτό να γίνει σε όλες τις χώρες και Ένωση και ΟΗΕ με καλύτερη ρωσινισμό από τώρα σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους. Δεύτερον, όσον αφορά τους περιφερειακούς οργανισμούς, και αυτό είναι μεγάλη καινοτομία, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, να έχουμε τέτοια συνεργασία, όπως με την Αφρικανική Ένωση συνειδητοποίησαμε ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και συμφέροντα, άρα το πιο λογικό είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, συνεργασία, εταιρική σχέση, Ξεκινήσαμε με το μεταναστευτικό, είπαμε να το χειριστούμε με σεβασμό και ανθρωπιά και να πάμε όμως τώρα και στην ανάπτυξη, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ασφάλεια και οπότε έχουμε πολλές δυνατότητες με συνεργασία τέτοια. Είναι η πιο βασική συνεργασία που μπορεί να αναπτύξει η Ένωση, Αφρικανική Ένωση. Έχουν αλλάξει νοοτροπίες και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Οι εκεί εταίροι μας εκτιμούν το έργο μας, για τα ανθρωπιστικά, για ειρήνευση, για ασφάλεια. Όμως αυτό που τους καίει σήμερα είναι επενδύσεις, θέσεις εργασίας, συνεργασίες σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και τελικά συνειδητοποίησαμε εμείς Ευρωπαίοι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά κοινά έργα, προγράμματα, κοινή δουλειά. Οπότε, αν είμαι καλά, πριν από τέσσερα χρόνια εδώ πέρασα την ακρόασή μου σε αυτή την αίθουσα πριν αναλάβω η πάτη εκπρόσωπος και όταν έφερα ως κορυφαία προτεραιότητα την Αφρική με κοίταξε ο κόσμος εδώ με πολλές επιφυλάξεις γιατί σκέφτηκαν ότι καλά γεωπολιτικά πρόκειται περί ανάπτυξης αυτό είναι η Αφρική και επιτρέψτε να είμαι λίγο κοινική ότι ακριβώς χάρη σε εισαγωγικά στην κρίση του μεταναστευτικού τώρα έχουμε ε, όλες αυτές τις παροχές τις αναπτυξιακές προς την Αφρική ξέρουμε πώς ήθελαν να επενδύσουν εκεί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί και σημαντικοί θεωρούν ότι η επένδυση είναι τρόπος να αποκτήσουν περισσότερη επιρροή, να εκμεταλλευθούν τους εκεί πόρους. Εμείς όμως λέμε ότι έτσι θωρακίζουμε τις κοινωνίες και είναι ευκαιρία και για τους νέους και για τις γυναίκες ε, που ανάπτυξη, εξέλιξη του ανθρώπου, ε, κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, δικαιώματα. Οπότε Γι' αυτό και κυρίως έτσι νομίζουμε ότι βοηθάμε τις τοπικές κοινωνίες να αποκτήσουν περισσότερη ποικιλία, ε, να προστατευτεί το περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι, τα διάφορα στάνταρ ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά τα εργασιακά. Να τι πάει να πει επένδυση. Γιατί έχουμε ειρηνευτικέ συμφωνίες, αλλά έτσι θα διαρκέσουν αυτές οι συμφωνίες, θα επιβιώσουν. Άρα αυτή η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης είναι το πιο βασικό. Εκεί επί τόπου έχουμε, είπαμε, μπούσουλα που είναι η συνεργασία με φορείς, με χώρες επιμέρους. Το 90% σχεδόν της εργασίας μας έχει διέπεται από προτεραιότητε που θέτουν οι εταίροι. Άρα αυτό το αναβαθμίζουμε περισσότερο και θέτουμε στον νέο προορισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κίνητρο τόσο ώστε να μπαίνουν στα προγράμματα οι τοπικοί μα εταίροι και αυτό θα είναι ο κανόνα τώρα. Αντισιακή συνεργασία για του στόχου βιωσιμή ανάπτυξη, την συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τον προπολογισμό, ε, είπαμε να έχουμε 30% προπολογισμό υυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο αφορά την εξωτερική μας δράση. Η μερίδα του Λέοντος η Αφρική, 30% περισσότερο. Τώρα την εποχή του Brexit και της λιτότητας καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για επανάσταση. Δεν είναι απλώς πρόοδος θετική, είναι επανάσταση. Τώρα όλα αυτά θα περάσουν από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Μην βιαστείτε, αλλά αποφασίστε το σωστό. Αυτό έχω να πω είναι η πρόταση που εμείς υποβάλλουμε, οπότε φυσικά και εμείς θα την υποστηρίξουμε. Μπίλα, μα θες, πες και εσύ δύο λόγια. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι αυτό χρειάζεται με το παραπάνω. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε. Είναι, είναι ο μόνος τομέας που κάνουμε τη διαφορά ως Ένωση, διότι πρόκειται για 20 δις κάθε χρόνο μόνο για την Αφρική. Ε, αυτό αυτό σας δείχνει το ότι εμείς και όχι καμία χώρα μόνη δεν μπορεί να καταφέρει. Είπαμε συνεργασία με ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνουμε ότι ποτέ το δημόσιο, το κράτος δεν μπορεί να αρκεί για τους στόχους βιωσιμής ανάπτυξης, γι' αυτό είναι το ειδικό τομέα, γι' αυτό θα μοντernίσουμε νέους τρόπους για κίνητρα, ούτως ώστε οι ιδιώτες να μπουν στο παιχνίδι των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Δύο παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα το εξωτερικό πρόγραμμα επενδύσεων για Αφρική και για την περιοχή γειτονία, να ελκύσουμε του ιδιώτε εκεί που χρειάζεται η επένδυση, που είναι η πιο ευάλωτη και εκεί που βέβαια είναι το πιο δύσκολο να γίνει η επένδυση γιατί υπάρχει γραφειοκρατία, δεν υπάρχει ασφάλεια, όλοι αυτοί οι διάφοροι τοπικοί διάβλοι της διοίκησης δεν υπάρχουν καν πρεσβείε σε πολλές χώρες. Όμως υπάρχουν παντού στην Αφρική αντιπροσωπείε τη Ένωση. Άρα έτσι μπορούμε να πλαισιώσουμε την προσπάθεια και έτσι να διευκολύνουμε τους ιδιώτες εκεί που χρειάζεται περισσότερα. Ιδιωτικές επενδύσεις που όμως συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Αν υπάρχει ψηλός κίνδυνος, ε, τότε έχουμε τα χρήματά μας ως εγγύηση για την επένδυση ακόμα είναι νωρίς, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε για το στόχο μας να πιστατεύουμε 44 δις μέχρι το 2020. Πολλά λεφτά. Επίσης διερευνούμε πώς μπορούμε να έχουμε εταιρείε τεχνολογίας. Ε, η Microsoft φυσικά είναι στο παιχνίδι και ένα από τα πρώτα προγράμματα αφορά το πώς θα υπάρξουν ψηφιακές δεξιότητες στους νέους της Τινησίας. Πολύ φιλόδοξο. Να το κάνει μόνο μία κυβέρνηση, αλλά είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν και οι ιδιώτες μόνοι τους χωρίς το δημόσιο. Είπαμε, εταιρείε τεχνολογίας για τους νέους Τινήσιους. Θεωρούμε ότι αυτό το πετύχουμε τα μέσα χρόνια. Σκεφτείτε τι δυνατότητες επιφυλάσσει το μέλλον. Φαντάζομαι από εδώ που θα σταματήσω θα ξεκινήσει ο Μπιλ. Έχουμε επίγνωση της ε, ευθύνης μας, ξέρουμε τα ωριά μας, ξέρουμε το πόσα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά, αλλά αν κανείς ε, βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των εταίρων μας, τότε καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο είναι το έργο μας. Ε, σας ευχαριστώ σε αυτή την υπέροχη αίθουσα και όσους ε, δουλεύουν στα θεσμικά όργανα και όσους όχι. Οπότε σας παρακαλώ όλους και τους μένει και τους δεν να κάνετε ό,τι μπορείτε και να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Να κάνετε ό,τι μπορείτε. Να επενδύσουμε σωστά στην ε, ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Πριν δώσω το λόγο στον Μπίλα, έχω το προνόμιο εγώ να μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, αλλά ξέρω ότι πολλοί άλλοι θα ήθελαν να σας θέσουν ερωτήσεις και μπορούν να αρχίσουν να γράφουν τις ερωτήσεις τους. Με πείσατε πάντως και νομίζω ότι όλους μας πείσατε Πραγματικά είναι πάρα πολύ πολύτιμο να έχουμε εσάς σε αυτή τη στρατηγική θέση. Εμπνέετε και υγείστε, αλλά στον, καλό, στον κακό μάλλον κόσμο εκεί έξω. Κάποιες φορές φαντάζομαι ότι το επιχείρημα αυτό είναι δύσκολο να το περάσετε. Εσείς επισκέφτεστε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συζητείτε με διάφορες ομάδες και φορείς. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που πιστεύετε πρέπει να αντιμετωπίσουμε εν ώψη και των ευρωεκλογών. Κυρία Μαγκέρνιν, θα είμαι μη ορθή ε, πολιτικός ε, και θα τα πω ντόμπρα όπως ε, συνηθίζω να κάνω. Έχω ξαναπεί ότι η μεταναστευτική κρίση άνοιξε το λέω με κινησμό, ένα παράθυρο ευκαιρίας για την αναπτυξιακή συνεργασία. Σε τεφά τον κακό κόσμο. Δεν είναι και τόσο κακός, απλά εστιάζει αλλού. Ίσως, τέλος πάντων. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αυτό είναι το επιχείρημα. Μην ξεχνάμε τι γινόταν πριν πέντε χρόνια ή δύο-τρία χρόνια πριν. Πού βρισκόμασταν τότε όταν όλοι είχαμε καταληφθεί από πανικό με τις ε, ε, μεταναστευτικές αυτές πιέσεις, με τα νούμερα των αφήξεων. Τα βασικά αίτια της μετανάστευσης ποια είναι. Είναι η έλλειψη ανάπτυξης, είναι η υγεία, είναι οι πανδημίες, είναι η αλλαγή του κλίματος οι συγκρούσεις, οι κρίσεις και όλα αυτά απαιτούν μακροχρόνιες επενδύσεις. Σήμερα από το διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου από το 85% το 85% έχει μειωθεί των αφήξεων και ίσως κάποιοι έχουν ξεχάσει τι γινόταν πριν από 2-3 χρόνια και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να πούμε ότι τώρα μειώνουμε τις επενδύσεις μας, ε, τα βασικά αίτια δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε πια γιατί σε 2-3 χρόνια θα έχουμε ξαναγυρίσει στην προτέρα κατάσταση, πριν από 2-3 χρόνια δηλαδή εκεί που βρισκόμασταν. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα, λόγοι που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ανάπτυξη. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό θα έλεγα σε εμά, αλλά στον κακό έξω, ε, κόσμο έξω θα έλεγα επενδύσει. Επενδύσεις που θα γίνουν θα είναι για την ε, ανθρώπινη εξέλιξη, για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Ε, αυτός είναι ο καλύτερο τρόπο. Και δεν μιλάω μόνο για την Αφρική, μιλάω για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να έχουμε ένα πιο ασφαλή κόσμο και μια πιο ασφαλή Ευρώπη. Θα επανέλθουμε ε, στους νόμους διαδρόμους, ε, μετανάστευση και τα λοιπά, αλλά αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να ε, δώσω τον μπαλάκι στον Μπιλ. Θέλουμε να προωθήσουμε αυτά τα παραδείγματα σαν το Ίδρυμα του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς που είναι πραγματικά σύμβολα του πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά ε, γιατί είναι πολύ καλή αυτή η συνεδρία και χαίρομαι για αυτή την αθρώα προσέλευση και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η φίλη Φεντερίκα Μογκερίνη. Σίγουρα η Ευρώπη υποτιμά τη σημασία ε, του έργου που έχει κάνει, τον ηγετικό ρόλο που έχει δείξει στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, με τα κονδύλια που αφιερώνει, κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και τους επόμενους μήνες θα αποφασίσετε αν θα αυξήσετε αυτή τη συνεισφορά στο τομέα 6 του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και κυρίως σε αυτά που κάνουμε εμείς ε, στα θέματα της ε, ανάπτυξης ε, και της κοινωνικής συμμετοχής. Ε, σε ό,τι αφορά το υπόβαθρο, στην πρώτη συνεδρία, στην επίσημη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε το 1958, τότε ήμουνα τριών ετών, το 1958 ήταν η χρονιά που ξέσπασε ο Μέγας Λιμός, που σάρωσε την Κίνα ε, και θέρισε τη ζωή δεκάδων εκατομμύριων ανθρώπων. Τότε το μέσο προσδόκιμο ε, όριο ε, στον κόσμο μειώθηκε κατά ένα χρόνο λόγω αυτού του λοιμού της Κίνας. Σήμερα η Κίνα και ο κόσμος είναι πολύ καλύτερα. Το προσδόκιμο ζωής τους είναι 77 χρόνια στην Κίνα, λίγο πάνω από το παγκόσμιο μεσόρο και μόνο 1% του κινέζικου του πληθυσμού μένει διαβεί σε όρους ακραίας φτώχειας. Και σίγουρα η Κίνα έχει σημειώσει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη, αλλά δεν είναι η μόνη χώρα που έχει αναπτυχθεί αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες. Το 1958 η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού διαβιούσε σε ακραία φτώχεια. Το 1958 ήταν 36%, σήμερα κάτω του 10% είναι οι άνθρωποι που ζουν σε ακραία φτώχεια. η αγαπημένη μου στατιστική πληροφορία και που είναι και ενδεικτικό του πόσο φροντίζει φροντίζουν οι άνθρωποι, τους συνανθρώπους τους, είναι η παιδική θνησιμότητα. Το 1990, 11 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν πριν την ηλικία των 5 ετών. Αυτό τώρα έχει μειωθεί στα 5 εκατομμύρια. Και παρόλο που ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί, έχει υποδιπλασιαστεί αυτή η παιδική θνησιμότητα. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ε, γενναιοδορία της ε, αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά και στην ε, ε, πρόοδο της επιστήμης, της ιατρικής και στην αύξηση του εμβολιασμού. Και σίγουρα υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας φτώχειας και της ε, γενεοδορίας στα αναπτυξιακά θέματα. Και σίγουρα η Ευρώπη είναι απαραίτητος εταίρος σε αυτή την αναπτυξιακή συνεργασία. Και παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 22% της παγκόσμιας οικονομίας, αντιπροσωπεύει το 57% της παγκόσμιας βοήθειας. Και ακόμη και δούμε τις δωρεές επίπεδο χώρας, μόνο τα κοινοτικά θεσμικά όργανα φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τέταρτη θέση με 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ να επενδύονται κάθε χρόνο στην αναπτυξιακή βοήθεια. Και βλέπετε με αυτή τη γραφική παράσταση στο κόκκινο τις ευρωπαϊκές δωρεές. Μετά βλέπετε το πορτοκαλί της αμερικάνικες δωρές και ως τμήμα της οικονομίας οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο γενναιόδωρες όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρά το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και δεν είναι υπέρ της εξωτερικής βοήθειας, παρόλα αυτά η Ευρώπη παραμένει γενναιόδωρη και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί Βέβαια το Κογκρέσο θα έχει ευτυχώ τελικά ε, τον τελικό λόγο για τον προσδιορισμό ε, τα, των επιπέδων αναπτυξιακής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ συχνά πηγαίνω επί τόπου και βλέπω πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια και η ποιότητα της αξιοποίησης των κονδυλίων σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως ε, στον τομέα της υγείας, που είναι αυτός που γνωρίζω καλύτερα, έχει βελτιωθεί αισθητά. Και η Παγκόσμια Συμμαχία για τον εμβολιασμό αξιοποίησε τις δωρές, ώστε τα σημαντικά αυτά εμβόλια που δόθηκαν στα παιδιά ε, μεσαίου εισοδήματο ε, στι εύπορε χώρε και στι αναπτυσσόμενε χώρε που κινδύνευαν να πεθάνουν από πνευμονία ή διάρρεια έχει γίνει χάρη στη συμμετοχή ε, της, της συνεισφοράς της ε, παγκόσμιας αυτής ε, του Ταμείου για, την παγκόσμια, για τον παγκόσμιο εμβολιασμό. Επίσης και το παγκόσμιο, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Εξάλληψη της Πολιομελίτιδας. Ξεκίνησε το 88 με 350.000 κρούσματα και σήμερα έχουμε 22 και προσβλέπουμε να εκμηδενήσουμε την πολιομελίτιδα. Και μάλιστα ήταν σημαντική η συνεισφορά της Ευρώπης ε, σε αυτή την προσπάθεια εξάλληψης ε, της πολιομελίτιδας. Και έχουμε και τα θέματα του Παγκόσμιου Ταμείου για την ε, καταπολέμηση ελονοσίας, φημασίωσης και AIDS, που έχει στοιχεί στη ζωή σε 120 εκατομμύρια. Και κάτι που δεν συζητάτε συχνά είναι πόσο σημαντική είναι αυτή η γενεοδορία που συμβάλλει στη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και στη μείωση των ασθενειών που μερικές φορές είναι απόρρια αυτής της φτώχειας. Και να δούμε πού θα οδεύσουμε προς τα που θα οδεύσουμε στο μέλλον και αν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρόοδο, μειώνοντας τη φτώχεια και βελτιώνοντας την υγεία. Εγώ είμαι αισιόδοξο γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος θα παραμείνει γενναιόδωρος και θα φέρουμε στο παιχνίδι και την καινοτομία. Πάντω οι προκλήσει είναι τεράστιε. και ένα από του λόγου που υπάρχουν αυτέ οι τεράστιες προκλήσει είναι η δημογραφική κατάσταση ε, των χωρών που γεννιούνται τα παιδιά. Και βλέπετε εδώ μια γραφική παράσταση που δείχνει ότι έχουμε 141 εκατομμύρια το χρόνο και έχει αυξη... αυξηθεί, ενώ θα μειωθεί στην υπόλοιπο τμήμα και μετά θα ανέβει. Αυτό που φαίνεται στο μπλε όμως είναι ότι οι γεννήσεις ε, εκτός της ε, υποσαχάριας Αφρικής, το κίτρινο είναι η υποσαχάρια Αφρική, σήμερα είναι 25% του συνόλου των γεννήσεων ενώ κατά τα υπόλοιπα αιώνα θα μειωθούν στο μισό. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ποσαχάρη Αφρική αντισταθμίζει το υπόλοιπο κόσμο. Γιατί εκεί στον υπόλοιπο κόσμο είχαμε από 104 εκατομμύρια μείωση στα 72 εκατομμύρια, ενώ η Ποσαχάρη Αφρική αυξάνει τι γεννήσει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μέχρι το 2050 90% των ανθρώπων που θα βρίσκονται σε ακραία φτώχεια θα μένουν στην υποσαχάριο Αφρική. Αυτή είναι η παρακαταθήκη και των υπόλοιπων χωρών και της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης των ασιατικών χωρών. Και αν φτάσουμε στο 2040, δεν θα είναι μόνο η Αφρική, αλλά η Νιγηρία, το Κονγκό θα έχουν πάνω από το 40% των πανφτωχων στον κόσμο και οι δύο αυτές χώρες θα έχουν ένα πληθυσμό 600 εκατομμυρίων. Δηλαδή οι δύο χώρες μαζί ε, θα έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καλά νέα είναι βέβαια ότι με τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην υγεία, στην παιδεία, ε, αυτή η δημογραφική αύξηση θα μπορεί να είναι στοιχείο θετικό, στοιχείο καινοτομία, μεγάλη απασχόληση και να οδηγήσει οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική. Το θέμα είναι θα διδαχθούμε από την Αφρική και η Κίνα και η Ινδία και θα εφαρμόσουμε αυτά τα διδάγματα κάνοντας επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και εδώ βλέπουμε τα διάφορα σενάρια για το πώς επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Αφρική. Και ποια θα είναι η συνέπεια. Αν ε, παραμείνουμε ισχυροί στις επενδύσεις, μπορούμε να οδηγήσουμε σε οικονομική ανάπτυξη, γιατί αυτή η νέα, η γενιά θα είναι πηγή παραγωγικότητας. Αν όμως δεν κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, τότε θα έχουμε υπαναχώρηση. Το ίδιο ισχύει και στην υγεία, με τον ιό του AIDS και την επιδημία του AIDS. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε με τη γενεοδορία μας ε, και να επενδύσουμε στα, στις νέες ε, τεχνικές για να μειώσουμε το AIDS. Θα σας μιλήσω λίγο και για την καινοτομία, γιατί ε, έρχομαι από μια διάσκεψη στο Βερολίνο που επιστήμονες από όλο τον κόσμο μιλούσαν για τα εμβόλια και τα νέα φάρμακα. Και είχαμε δοκιμές για ένα νέο ε, εμβόλιο φυματίωση. Ε, θα χρειαστούν βέβαια χρόνια για να το αναπτύξουμε και να, το, και να κυκλοφορήσει. Θα μειώσει όμω αισθητά του θανάτου από φυματίωση. Και δεν μιλούμε μόνο για τη φυματίωση. Δεν έχουμε μόνο στα θέματα τη φυματίωση και ανοτομία και στα εμβόλια. Αλλάζει ο τρόπο ε, παρασκευή των εμβολίων. Έχουμε τα εμβόλια που στηρίζονται στον αγγελιοφόρο RNA. Και πολλέ εταιρείε όπω η CureVac AG ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Θα αλλάξει ο τρόπο που θα παρασκευάζουμε τα εμβόλια. Και σε λίγους μήνες και όχι σε 3,5 χρόνια που είναι κατά μέσο όρο ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός εμβολίου θα κάνουμε στο μέλλον τα εμβόλια χάρη στη χρησιμοποίηση του Ευαγγελιοφόρου RNA και γι' αυτό χρειάζεται αύξηση του προϋπολογισμού επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας αλλά και του προϋπολογισμού για την έρευνα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε τα εργαλεία ώστε να αποκτούν οι γεωργοί καλύτερους σπόρους και να αποφεύγουν τις ε, ζημιές από τις κλιματικές αλλαγές και τις ακραίες καιρικέ συνθήκες. Ε, και αυτό θα το καταφέρουμε και χάρη στην καινοτομία, γιατί οι κλιματικές αλλαγές είναι υπαρκτές ε, και είναι τεράστια η πρόκληση και για την καινοτομία για να αποφύγουμε τα καυσαέρια και τα αέρα του θερμοκηπίου και η γεωργία της επιβίωσης στην Αφρική να μην γίνει το εξηλαστήριο θύμα των κλιματικών αλλαγών γιατί τελευταία πενταετία δεν είχαν καλές ε, σοδιές. Θα πρέπει λοιπόν πολλά να γίνουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Και γι' αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί ο ηγετικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά. Και όλε οι υπόλοιπε χώρε και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να κρατήσουν ε, τι ε, υποσχέσει του. Πρέπει να είστε υπερήφανοι για τη γενναιοδορία σα και Ελπίζω να κρατήσετε αμύωτη την καινοδορία σας και στην επόμενη επταετία και να την φέρετε σε ένα νέο επίπεδο. Ευχαριστώ. Πόσο ωραία να έρχονται κάποιοι στο σπίτι σου και να σε εγκομιάζουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπίλ, γιατί μας έβαλες στο σωστό μονοπάτι για το μέλλον. Το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας σου, Μπιλ, είναι πώς ε, διατάραξες ε, ε, τον κόσμο μέχρι τώρα, εσύ και ο Πολ Άλλαν, με την εφεύρεση του προσωπικού υπολογιστή. Η αλλαγή του κλίματος, πιστεύεις, θα δημιουργήσει αντίστοιχο αριθμό τιμένων νικητών και αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Είναι ηρωνία το ότι οι υπεύθυνοι για την αλλαγή του κλίματος, οι πιο εύπορες χώρες δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια εκπέμπουν ε, τις, ε, τους ρήπους και δεν έχουν ε, υποφέρει τόσο. Σίγουρα υπήρξαν καύσονες, υπήρξαν διάφορα ακραία φυσικά φαινόμενα, όμως ο δραματικός αντίκτυπος θα είναι αλλού θα είναι στο Ισημερινό και στις φτωχές περιοχές. Πρώτα απ' όλα στην Αφρική, που δεν έχουν κάνει και τίποτα οι άνθρωποι για να προκαλέσουν τέτοια αλλαγή του κλίματος. Μεγάλη αδικία. Ε, κάποιοι θεωρούν ότι η αλλαγή του κλίματος δεν είναι πρόβλημα και αυτό πραγματικά πονάει. Ε, κάποιοι λένε ότι η αιωλική ηλιακή ενέργεια είναι φθηνέ πηγές ενέργειας και έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Ούτε αυτό βοηθάει όμως, γιατί ε, πρέπει να κάνουμε ευρύτατες αλλαγέ και χρειαζόμαστε αξιόπιστες πηγέ ενέργεια, πρέπει να αλλάξουν μεταφορέ, συγκοινωνίε, όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά τα πάντα. Σιδηρόδρομοι, αεροπλάνα, φορτηγά, χαλιβουργία, λιπάσματα, τσιμέντο, όλα πρέπει να αλλάξουν. Η ε, θέρμανση των κτηρίων και ούτω καθεξής. Επομένως, ε, ε, στον τομέα της καινοτομίας και εκεί πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Σήμερα με τον Επίτροπο Μοέδας αναγνώρισα ότι υπάρχει ένα, ε, μια συγκέντρωση πόρων από ένα ίδρυμα το οποίο προεδρεύω για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας. Άρα υπάρχει δράση. Τώρα, κατά πόσον αυτό κινείται με γρήγορους ρυθμούς ή όχι, δεν ξέρω. Σίγουρα ε, θα έχουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι το σενάριο, 1,5 βαθμός Κελσίου, 2, ε, αλλά και να καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλά επίπεδα, θα έχουμε πολλά προβλήματα ε, και υπάρχει και η Επιτροπή για την Προσαρμογή. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν στο μέτωπο του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να μην σχετίζονται μεταξύ τους. Για τα φωτοβολταϊκά, για την Αφρική, μα έχουν 2% των εκπομπών. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα να βάλουν φωτοβολταϊκά ε, οι Αφρικανοί. Ναι, φυσικά καλό θα ήταν να το κάνουν, είναι και φθηνότερο το σύστημα αυτό, αλλά οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπο κόσμος, κυρίως ε, οι χώρες μεσοεισοδήματο, η Κίνα ε, πρώτη που θα πρέπει να προβούν στι αλλαγέ αυτές. Είναι όλα συναρπαστικά, αλλά σίγουρα φοβίζουν. Πρέπει να δούμε, θα κάνουμε συλλογικά αυτό που πρέπει. Για μένα Δύο είναι τα προβλήματα που ζητούν παγκόσμια δράση. Το πρώτο είναι η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να συνεργαστούν οι χώρες γιατί από μόνες τους δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά και οι πανδημίες όπως η γρήπη ε, δεν ε, ε, επηρεάζουν με τη όλο το πλανήτη. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των χωρών για την αποφυγή πανδημιών Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για μένα τουλάχιστον και μόνο με συνεργασία μπορούν να επιληθούν. Ναι, συζητήσαμε το πρόβλημα με τους ανθρακορίχους και στη χώρα μου και στη δική σου και σε πολλές άλλες χώρες. Πώς θα βοηθήσουμε να υπάρξει αυτή η μετατόπιση ανώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Μέχρι τις, 10, μέχρι τις 5 και 10 λέει ένα σημείωμα που μου βάλαν μπροστά μου. Ναι, το σημείωμα τα λέει αυτά, λέει κύριε Τέλος πάντων, λοιπόν, Παρακαλώ, έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση. 90 δευτερόλεπτα θα έχει όποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση. Θα δούμε πόσος ε, χρόνος μένει. Εσείς πρώτα και μετά η κυρία στο βάθος. Παρακαλώ, εσείς 90 δευτερόλεπτα. Λιγότερα μου φτάνουν. Άρνε Λίτς λέγομαι και είμαι ευρωβουλευτής από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Η Φεντερίκα Μογκερίνη είπε κάτι και εμεί είμαστε υπέρμαχοι ω σοσιαλιστέ δημοκράτε, υπέρμαχοι των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, ότι θέλουμε να προωθήσουμε την προοδευτική κοινωνία. Εσεί ε, τι πιστεύετε, είναι έτοιμη η ευρωπαϊκή κοινωνία να προωθήσει του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τη συζήτηση αυτή, να μπει στο προσκήνιο δηλαδή, να είναι ένα πλαίσιο για τι ε, συζητήσει που θα έχουμε. Είπατε πολλά πράγματα και εσείς για την ηλιακή ενέργεια, την Αφρική κτλ. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτό το θέμα στην πολιτική γενικά και όχι μόνο εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, ωραίε είναι ερωτήσει. Καλό είναι και να υπάρχει μια συμβουλή, συμβολή στη συζήτηση. Εξίσου καλό και αυτό, Φροντζούλικα. Ευχαριστώ η σχέση μεταξύ τεχνολογία και στόχων βιώσιμη ανάπτυξη είναι στον πυρήνα κάποιων συζητήσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί ότι και η ψηφιακή τεχνολογία έχει ένα μεγάλο δυναμικό για την επίτευξη αυτών των στόχων, όμως έχουμε και κάτι άλλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις αναψώμενε χώρες ιδιαίτερα, αυξάνοντας τις ανισότητες και δημιουργώντας αρνητικές ε, εξωτερικές επιπτώσεις. Πολλά είναι τα ωφέλη από τεχνολογία, αλλά υπάρχουν και 3,5 δις άνθρωποι που δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Επομένω, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καινοτομία να μην διωγγώσει το χάσμα που ήδη υπάρχει στην κοινωνία μεταξύ αυτών που ωφελούνται από την πρόοδο τεχνολογία και αυτών που δεν ωφελούνται. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις χωρίς όμως ε, την καινοτομία για την οποία κάνατε λόγο κύριε Γκέιτς, κυρία Μογκερίνη να την ε, καταστήλουμε γιατί αυτή οδηγεί στην ε, ανάπτυξη. Υπάρχουν και τρει βουλευτέ, λέει ο Σάιμον, αλλά θέλω να ακούσουμε και φωνέ ανθρώπων που δεν είναι ευρωβουλευτέ. Ε, σύντομα, εσεί πίσω στο βάθο. Η Ελιζαμπέτα. Και κλείνει το μικρόφωνο τη. Α, είμαι εκπαιδευόμενη. Μαθητευόμενη μάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλές φορές επεκρίνεται η Ένωση. Και ξανασβήνει το μικρόφωνο. Για το τι γίνεται όταν δίνει κάποιες ενισχύσεις σε σχέση με τη, τη, τους και στα Βαλκάνια έχουν υπάρξει κινήματα κατά των εμβολίων. Αυτό όμως δεν είναι κίνδυνος και υπάρχουν και οι αυτοάνωσες ε, ασθένειες, λύσουν τα παιδιά. Τι γίνεται με την πολιτική αυτή των εμβολίων. My name is Antonella, I'm director of Young Water Solutions. Um, we empower young people to become entrepreneurs. Θέλουμε να φέρουμε την επιχειρηματικά των νέων και ακούσαμε για κάποια νέα από την Ρουάντα, 22 ετών, να μας πει Μα είπε τι γίνεται. Τι, εσείς τι λέτε για γερμογερίνη, τι, τι λέτε, πώ γίνεται να γίνουν επιχειρηματίε, να φτιάξουν κάποιε κοινωνικέ επιχειρήσει και να βοηθήσουν στόχου. Καλύτερα προτάσει θέλω και όχι ερωτήσει, Μα Μίκινς. Προ τον κύριο Γκέιτ από την Λετωνία. Έχουμε φιλοσοφική, ακούγεται η ερώτηση. Πώ βλέπετε τον κόσμο, πώ βλέπετε τον πολιτισμό την επόμενη πεντηκονταετία, πόλεμοι, τεχνολογία, ο ρόλος Ευρώπης δηλαδή. Κύριε Κούλογλου. Mr. Gates, uh, um, my name is Στέλιος Κούλογλου. Στέλιος ονομάζομαι κύριε Gates και είμαι ευρωβουλευτής από την πολιτική ομάδα της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με εφετηρία την οικονομική βοήθεια προς τις ενδεξόμενες χώρες μέχρι και την υπόθεση αλλαγής του κλίματος. Η κυβέρνηση Τραμπ ε, έχει υιοθετήσει μάλλον αρνητική θέση, λιγότερο θετική τέλος πάντων από την θέση της Ένωσης. Πώς το βλέπετε αυτό? Δεν μπορούμε να βρούμε, δεν μπορείτε εσείς να βρείτε ε, κάποιο είδους λύση συνεννόησης με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο επόμενος κύριος, ο κύριος Πόπα. Πώς λέτε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, ιδίω που ασχολούνται με τα ψηφιακά, να φορολογηθούν εκεί που δημιουργούν τα κέρδη τους και όχι εκεί που είναι η έδρα τους. Σάιμον, έχουμε 9 λεπτά και σας είπα προηγουμένως ότι πολλές φορές δεν μπορεί να βρει λύση για όλα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως για απάντηση για κάθε θέμα ανάπτυξη είναι το ETTG. Για πέστε μας. Uh, Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Μαγκερνή και τον κύριο Γκέιτς γιατί αν κάποιος είναι σε θέση να μιλάει για νεοδορία είστε κατεξοχήν εσείς. Και το να μιλούμε για την ανανεωμένη εταιρική σχέση, ε, αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και σίγουρα αυτά τα δύο θέματα είναι αλληλένδετα, γιατί η γενοδορία και η εταιρική σχέση είναι έννοιες ε, που εντάσσονται στην άποψη ότι η συνεργασία είναι η καλύτερη προσέγγιση για να επιληθούν προβλήματα και να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις, ε, ξεπερνώντας τα σύνορα και δε, χωρίς να βάζουμε πρώτα τα συμφέροντά μας. Γιατί τα συμφέροντα μερικές φορές είναι ε, ένα σύντομο δρόμος ε, του, της ιδέας ότι προηγούνται τα δικά μου συμφέροντα από τα δικά σου συμφέροντα. Το θέμα είναι να βρούμε τα κοινά σημεία και τα κοινά μας συμφέροντα. Και νομίζω ότι αυτά που είπατε ε, συμβάλλουν ε, σε αυτό και η δική μας οργάνωση, η TDG, εντόπισε το τομεί όπου σε ορισμένα θέματα μπορούμε να βρούμε απαντήσεις και έτσι μπορούμε να κάνουμε την επανάσταση της βιωσιμότητας, να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να προσαρμοστούμε σε αυτές, να κάνουμε δίκαιη την παγκοσμιοποίηση και φτάνουμε και στο θέμα της ψηφιοποίησης, γιατί η Κίνα πολύ αποτελεσματικά μείωσε τη φτώχεια και αναπτύχθηκε οικονομικά, αλλά με όρους που έχουν αλλάξει σήμερα και η πρόοδος της ψηφιοποίησης και της τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τους όρους. Θα χρειαστούν νέοι κανονισμοί για την ρύθμιση και για την προσαρμογή στην ψηφιοποίηση και να δώσουμε και σε, σε ανθρώπους που δεν έχουν τις ψηφιακές δεξιότητες να ζήσουν σε αυτή την ψηφιοποιημένη οικονομία. Επίσης, οικοδόμηση της ειρήνης, αποτροπή πρόληψη των συγκρούσεων. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμέλια της διεθνούς συνεργασίας, της πολυμέρης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικές φορές υπάρχει αντίληψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η πολυμερή συνεργασία είναι ε, σχέδιο των ελίτ και όχι του κοινού. Και σίγουρα εκεί έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε αλλά όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, γιατί δεν μπορεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκαταστήσει την έλλειψη δράση και δέσμευση υπέρ τη κοινωνική δικαιοσύνη των κρατών μελών. Και όσοι ενδιαφέρονται για τη διεθνή συνεργασία, το βιώσετε κι εσεί ε, στο Ίδρυμά σα, κύριε Bill Gates. Αν δεν βρείτε του κατάλληλου εταίρου, οι προσπάθειε σα ε, είναι μάτε. Και το νιώσαμε κι εμεί αυτό στην αναπτυξιακή συνεργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι με την ψηφιοποίηση θα πρέπει να επενδύσουμε στην κατανόηση της ψηφιοποίησης τεχνολογικά και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για τις χώρες που έχουν διαφορετικά συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και νομίζω ότι το θεμελιώδες ερώτημα εδώ είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ε, να εποφελείται το κοινό, ο κόσμος και γι' αυτό το σημαντικό είναι τα φορολογικά συστήματα και έτσι σίγουρα είστε γενναιόδωρος και θέσει είναι καλύτερη. Αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ ακαθόδες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη να συμφωνήσουν σε ένα φορολογικό καθεστώ που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση των δημόσιων δράσεων που χρειάζονται για το κοινό καλό και στα κράτη μας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περιφερειακό επίπεδο σίγουρα οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και το θεματολόγιο του 2030 είναι μια ενθάρρυνση για πολιτικές που θα εξυπηρετούν το κοινό καλό σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι ε, η άγουσα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να προσχωρήσουν αυτό και τα κράτη-μέλη. Χαίρομαι πάντω που αν μη τι άλλο σε αυτή την αίθουσα υπάρχει συμφωνία. Και σίγουρα το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτέ τι πέντε δράσει, αυτού του πέντε άξονε και ε, ε, σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και επίσης είναι σημαντικά σημεία για την προεκλογική εκστρατεία ενώπιση των ευρωεκλογών. Και σίγουρα μπορεί να μην σα εξασφαλίσει τη νίκη βράχη πρόθεσμα, αλλά είναι σημαντικό να προγραμματίσουμε και μακροπρόθεσμα αυτή τη συζήτηση στις κοινωνίες μας. Αλλιώς θα την ξεχάσουμε και μερικές φορές ο βραχυπρόθεσμη εθνικιστική ερμηνεία και κοντόφθαλμη είναι αντιπαραγωγική. Και σίγουρα η εταιρική σχέση σχέση Ευρωπαϊκή Αφρικής είναι, θα είναι η λιδία λίθο αυτού τη νέα αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν θα πρέπει να επενδύουμε σε μονοπόλια το που υπάρχουν οι λύσει και που υπάρχουν τα προβλήματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού αυτά τα προβλήματα και να βρούμε κάποιου δρόμου και να αναζητήσουμε κοινέ λύσει. Ναι, ναι, το ξέρω. Τελεία. Στην τελευταία σύνοδο είπατε θα αναπτύξουμε, ε, θα εμβαθύνουμε ε, την ε, συνεργασία. Ο Μπίλ δύο λεπτά και πριν φύγει και η Φεντερίκα για να κλείσει. Και έπειτα θα συζητήσουμε εμείς με τους εισηγητές. Ο Μπίλ Γκέιτς. Έγιναν πολλά καλά σχόλια. Το φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πιο προοδευτικό ε, στις χώρες, κρατικοί φόροι, φόροι εταιριών. Δεν είμαι βέβαια ειδικό για καμία χώρα, ίσως πλην τον είπα. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν προοδευτικά συστήματα. Η ψηφιακή τεχνολογία σε, ως επιτοπλίστων είναι ευλογία, συνοδεύεται βέβαια από κάποιες προκλήσεις, ίσως και απρόβλεπτε ακόμα και για τους δημιουργούς ε, των νέων τεχνολογιών. Αλλά προσπαθούμε παραδείγματο χάρη να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία στην ε, Αφρική. Να υπάρχει ψηφιακέ ψηφιακές τραπεζικές συναλλαγές ε, με πολύ χαμηλά τέλη είναι όφελος αυτό. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί η κρατική απόδοση, οι κρατικές επιδόσεις να δούμε ας πούμε αν δίνονται επενδύσεις για το σχολείο. Παίρνεις μια φωτογραφία, τη στέλνεις. Είναι σχολείο αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία ή όχι. Αν όχι υπάρχουν και ούτω καθεξής. Σίγουρα ε, θα πρέπει να υπάρξει ε, αυτάρκεια και να μπορεί να τα ε, καταφέρνει από μόνη της η Αφρική και γι' αυτό προϋπόθεση είναι η κρατική δίκη να λειτουργεί σωστά. Όσο υπάρχει ε, γενεοδορία μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η συνολικά στη ΣΥΠΑ θα διατηρηθεί η πολιτική. Το Κογκρέσο έχει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο θα έλεγα και μια πιο υπεύθυνη άποψη θα μπορούσα να πω από ότι το εκτελεστικό σώμα αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση δηλαδή. Τώρα για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Υπάρχουν 17 στόχοι και πολλοί επιμέρους στόχοι. Εμείς τι κάνουμε. Ε, έχουμε τα λεγόμενα, τους λεγόμενους goalkeepers ε, και παρακολουθούμε πού υπάρχει καινοτομία, πού υπάρχει πρόοδος και επίσης πού υπάρχει υποχώρηση. Το βλέπουμε ρεαλιστικά. Λέμε κάποιοι στόχοι είναι πιο φιλόδοξοι, κάποιοι είναι πιο εφικτοί. Σίγουρα όλοι πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση και προσφέρουν νομιμοποίηση ως προς το τι θέλουν ε, οι χώρες κατά πολέμηση της πολιομιελίτιδας ε, και κρίζωση της νόσου εν τέλει όπως και του ιού του έτσι κτλ. κτλ. Βασικά αυτά είχα να πω ως απάντηση. Κυρία Μογκερίν, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είμαι στο ίδιο πάνελ με τον Μπίλ γιατί παίρνει όλες τις ερωτήσεις και δίνει και όλες τις απαντήσεις. Ε, τέλειο αυτό. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο είναι ότι η δημογραφική κατάσταση στην Αφρική είναι ακριβώς όπως περιέγραψε τα πράγματα ο Μπίλ και για μας τους Ευρωπαίους είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη συνεχώς ότι 17 χιλιόμετρα μακριά είναι η Αφρική από εμάς ε, και ε, επειδή είμαι από την Νότια Ευρώπη, αν πάει κανείς από την, ε, την Ισία στη Μάλτα, πάει νότια. Άρα είναι νότια Αφρική μέρος της Ευρώπης. Δεν είναι τα πράγματα ή άσπρο ή μαύρο, είμαστε όλοι μαζί εδώ. Αν αποτύχει η Ευρώπη, δεν πρόκειται να πετύχει η Ευρώπη. Ίσως κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι μπορεί να είναι πιο χαλαροί. Εγώ δεν το πιστεύω γιατί είμαστε παγκοσμιοποιημένοι. Αλλά η Αφρική σίγουρα είναι η γειτονιά μας για μας, την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να είναι γενναιόδορη και αυτό είναι ο πιο ευφύς τρόπος ε, να κοιτάμε το δικό μας συμφέρον, αν θέλετε. Ε, ο εγωισμός ε, έτσι θα φανεί, με τη γενναιοδορία. Δεύτερον, και τελευταίο. Ρώτησαν κάποιοι πώς ε, οι νέοι Αφρικανοί μπορούν να, ε, να αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα, πώς μπορούμε να τους ε, χειραφετήσουμε, να τους ενδυναμώσουμε. Θέλουμε να τους δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Τι σας λένε οι νέοι Αφρικανοί άνδρες και γυναίκες, πρόσβαση στην παιδεία, σε κονδύλια, καταπολέμηση της διαφθοράς, λογοδοσία, διαφάνεια, μια λογική γραφειοκρατία, υποδομές υλικές αλλά και ψηφιακές, πολύ σημαντικές ψηφιακές, να υπάρχουν σωστές και πρόσφαρες συνθήκες και μιλώ και για το κλίμα, κλιματική αλλαγή δηλαδή και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν αρκεί η ανάπτυξη, επενδύσεις, πρέπει να γίνουν σε όλους τους τομείς. Η έρευνα, εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και ο Μπίλεχ σωστά είπε για τον προπολογισμό. Επενδύουμε σε εξωτερικές δράσεις αλλά και σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η έρευνα. Γιατί αν κάνεις μόνο ένα πράγμα δεν το λύνεις το πρόβλημα ώστε να μην το λύσει τόσο άλλο το πρόβλημα, αλλά αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο ε, για να βρούμε σωστέ απαντήσει και να λύσουμε τα προβλήματα. Και τελευταίο σχόλιο, φαντάζομαι είστε πεπισμένοι όλοι όσοι είστε σε αυτή την αίθουσα, ε, ε, το θέμα είναι όμως ε, να πείσουμε τους υπόλοιπους ε, και σίγουρα αυτό είναι σημαντικό για τους ευρωβουλευτές που θα πρέπει να βρουν τις απαντήσεις και να διεξαγάγουν και μια προεκλογική εκστρατεία σε λίγο. Τους να πείσουν την ε, κοινή γνώμη. Χρειάζεται σθένος και θάρρος για να τεθούν κάποια ζητήματα σήμερα στην Ευρώπη. Και αυτό το σθένος πρέπει να το δείξουμε. την ώρα που μιλάμε, οι επενδύσεις στην ανάπτυξη έχουν νόημα. Είναι κάτι λογικό, είναι το φυσιολογικό που πρέπει να γίνει. Το ερώτημα είναι, θα κάνουμε το σωστό και το λογικό. Θα πάρουμε τις λογικές αποφάσεις, ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εμείς Ευρωπαίοι, έχουμε παραμείνει αρκετά λογικοί και η πρόκληση τώρα είναι ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας να συνεχίσουμε να είμαστε ε, και λογικοί αλλά και εγωιστικά γενναιόδοροι. Ευχαριστώ. We, we defend development, we Ναι, θέλουμε ανάπτυξη και τη συζητούμε και σε βάθος. Όλα αυτά είναι και στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ήσασταν πηγή έμπνευσης και σας ευχαριστούμε.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 If those were leaving, there's a way out here because we're going to start Παρακαλώ ποιος θέλει να αποχωρήσει ησύχως. Εκτός από την γαλαρία μπορείτε και από εδώ μπροστά να φύγετε. Ταχύτερα, λέει η πρόεδρος. Okay, we're going to... Μάξουελ, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το θέμα της ανάπτυξης, να το συζητήσουμε και εις βάθος όπως λέγαμε Έχουμε τώρα τον James Mackey, διευθυντής της ECDPM, μέλος της ETTG, ο Σεμπάστιαν Τρέιερ επίσης. Έχετε τον λόγο. Ο κύριος Μάκη πρώτος, πολύ ενδιαφέρον αυτό το απόγευμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Bill Gates και τη Φεντέργα Μογκερίνη που ήρθαν και αυτό που συνεκράτησαν πρώτα-πρώτα είναι αυτό που είπε αρχή-αρχή η Λίντα ότι ήρθε την πιο επίκαιρη στιγμή το θέμα. Ή τέλος πάντων τη στιγμή που είναι πιο επίκαιρο. Τώρα που πάμε για τις ευρωεκλογέ, για την καινούργια κομισιόν, άρα πολλά πρόκειται να κουβεντιαστούν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η φάση. Και εμείς ως ETTG, ως Think Tanks θα πρέπει να συμβάλλουμε. Πολύ σημαντικό πλαίσιο επομένω οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη για ε, Υπόσχεση προ την ανθρωπότητα. Το καλύτερο που έχω ακούσει. Η καλύτερη περιγραφή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Πάντω, χάνουν λίγο από τη λάμψη τους μέσα σε όλες τις τεχνοκρατικέ προσπάθειες που τι πλησιώνουν. Πάντω, συνεχίζουν να αποτελούν ένα πλαίσιο που θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε επίσης. Αυτό που μου έμεινε από σήμερα είναι ότι θα πρέπει να παραλυφθεί δράση. Κοινή δράση. Αυτό πάει να πει στο γεωσμής ανάπτυξης. Αλλά είδατε πόσες φορές επανελήφθη αυτή η διαβεβαίωση. Εταιρικές σχέσεις στην ανάπτυξη, σύμφωνα στην, στην αναπτυξιακή βοήθεια είναι αυτό κάτι ρευστό, αλλάζουν οι εταίρες. Και, κατά τρίτο λόγο, ο ίδιος ο Bill Gates τόνισε ότι αποδίδει αναπτυξιακή βοήθεια και αξίζει κανείς να ξοδεύει για αυτήν. Σώζονται σοές. Κατά τις φτώχειες, κατά τις αρρώστιες. Άρα κανείς έτσι δεν πρέπει να τα δει και μακρόπνο βλέπει την πρόοδο. Είπαμε θα πρέπει, όπως λέει το θέμα μας, ε, να είμαστε καινοτόμοι, να αλλάξουμε μεθοδολογία και κατόπιν όσων είπε ο κόσμος σήμερα δεν ξέρω. Είμαστε καινοτόμοι, έχουμε εξέβρει νέες λύσεις. Φυσικά και αφού αποδίδει αυτή η πολιτική να συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει να πασχίσουμε περισσότερο για καινοτομία. Τι Σιλίντα, μα είπες ότι πολλές φορές αφήνουμε απ' έξω από την κουβέντα τα πιο σημαντικά. Τα αποφεύγουμε τώρα, είπαμε ότι όλα αυτά δεν είναι νέα, αλλά είπαμε ότι η αναπτυξιακή αρρωγή δεν αρκεί, υπάρχουν και άλλα μέσα και άλλα εργαλεία, περισσότερα χρήματα κατά της φτώχειας, αλλά να αντιμετωπίσουμε και την αλλαγή του κλίματος και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και όλα αυτά απαιτούν χρήμα, συνέργειες, μέθοδοι, αποδοτικές. Λύσεις για όλο τον κόσμο που να αποδίδουν. Να δούμε επίση πω θα το δράσουμε και μέσα στην Ευρώπη και όχι μόνο εκτός αυτή. Γιατί βλέπω ότι δυσκολευόμαστε κάπω για το τι θα κάνουμε εδώ. Να δούμε πώ. θα αναπτύξουμε κάποιε πολιτικέ εδώ για το εσωτερικό. Και αυτό μας έχει προβληματίσει αρκετά Βέβαια όλοι εδώ είμαστε ειδικοί στην διεθνή πολιτική. Τώρα όσον αφορά το πώς μπορούν να βρεθούν νέες μέθοδοι δεν είναι μόνο τα τεχνικά, δεν είναι μόνο επιστημονικές επιτυχίες, ανακαλύψεις, είναι και θέμα διοίκησης, διαχείρισης, ότι δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουμε ε, να έχουμε με τη συνήθεια τις παλιές μεθόδους Βέβαια δεν έχουμε όλες τις λύσεις. Ίσως μπορούμε να εμπνευστούμε και από τους κατατόπους εταίρους στον υπόλοιπο κόσμο. Να δούμε που έχουμε κοινού παρανομαστές. Να μην αποφασίσει μόνο η Ευρώπη. Ποια είναι η λύση. Πολύ πολύ μιλητές το είπαν. Και εν κατακλείδη ο διάλογος με την Αφρική, το είπαμε, μία-δυο φορές ότι τελικά να δούμε τι θα πει κοινή πορεία, κοινή συνεργασία με τους Αφρικανούς, τις άλλες όχθες της Μεσογείου. Άρα αμφίδρομα να είναι τα πράγματα. Επίσης για το πολιτισμικό πλαίσιο μάλιστα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις τεχνικές, είναι τεχνολογικό το θέμα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, αλλά δεν είναι θέμα σχεδιασμού, είναι υπευθυνότητα, ευθύνη τη επόμενη Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με την λογοδοσία, τι ρόλο θα έχει η κοινωνία των πολιτών, αυτά. Η διερμηνία θα σταματήσει στις 5.30. Φαντάζομαι ότι παρά 20 και εμεί θα ολοκληρώσουμε. Σεμπάστιαν, ναι, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι στο πρώτο πάνελ Ακούσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και πρέπει να προωθήσουμε την ανάγκη επενδύσεων ε, ε, ότι δεν είναι μόνο για το δικό μας όφελος αλλά και για να προωθήσουμε και να ε, υπερασπιστούμε τις αξίες μας, πολυμέρεια, καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτές είναι οι αξίες πρέπει να περασπίσει η Ευρώπη. Βασικό στοιχείο. Επίσης, και στο, στις χώρες μας πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, είπε και ο Τζέιμς ότι η επίσημα αναπτυξιακή βοήθεια δεν αρκεί. Πρέπει να επενδύσουμε και στην παγκοσμιοποίηση, στο εμπόριο και πώς αυτά σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας και τις ανισότητες. Πρέπει και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. η νέα ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης και αυτό πρέπει να μπει στη, ψηλά στην ατζέντα. Και με τον Bill Gates η συζήτηση έδειξε ότι η καινοτομία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι μεγάλος κομμάτι του προπολογισμού του πολιτού μεσονικού πλαισίου πρέπει να πάει εκεί η καινοτομία στην Ευρώπη και σε συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους. Σημαντικά και αυτά. όχι απλά να μεταφέρουμε τη δική μας καινοτομία εκεί, αλλά να τους επιτρέψουμε ε, να δημιουργούν εκεί καινοτομία. Για το τελευταίο, ο Σάιμον έδωσε μεγάλη έμφαση στο ότι στρατηγική σημαίνει και επιλογές. Πολύ σωστά έδωσε έμφαση σε αυτό. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε έτσι. το είπε και η Νατάλη. Πρέπει να αυξήσουμε το ποσό, αλλά να κάνουμε και επιλογές. Μπορούμε να τα έχουμε όλα αν έχουμε ένα μακρό πνόρα. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε αν θα χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη ε, ή την ε, συνεργασία ή κάτι άλλο. Όχι. Πρέπει να τα επιλέξουμε. Λοιπόν, πριν χάσουμε τους δερμηνείς, ε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο τους. Εδώ η δερμία σταματά. Σας ευχαριστούμε.